Uh, Καλησπέρα σας αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα πρώτα να εγκρίνουμε την ημερήσια μας διάταξη. Ε, σήμερα, ημέρα Δευτέρα 18 Μαρτίου, η συνεδρίαση ε, θα διαρκέσει από τις 3 μέχρι τις 6.30. Ε, Επίσης, θα ακούσουμε επιπλέον ενημέρωση για το Ευρωπαϊκό Κέντρο Έρευνας και Εκανοτήτων Ασφάλειας στον Κυβερνοχώρο, μια και διεξήχθη στις 13 Μαρτίου στο Στρασβούργο σχετικός τριμερής διάλογος και μια επιπλέον ενημέρωση για τις ευρωπαϊκές στατιστικές ε, των επιχειρήσεων, μια και ο σχετικός τρίλογος έγινε στις 14 Μαρτίου στο Στρασβούργο. Με μάλιστα αίσια διεκπαιρέωση της συμφωνίας εκ μέρου τη διαπραγματεύτική μα ομάδα. Αν δεν υπάρχουν άλλα σχόλια, θα ήθελα να εγκρίνουμε παρακαλώ την ημερήσια διάταξη. Δεν βλέπω άλλα σχόλια, ούτε κι εγώ έχω συγκεκριμένε ανακοινώσει, οπότε μπορούμε να περάσουμε στο σημείο 3 τη ημερήσια διάταξη. τη μελέτη για το πώ μπορεί να ενισχυθεί η σύζευξη τομέων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να προωθηθεί η σταθερότητα του δικτύου και η υπαλλαγή από τι εκπομπέ διοξιδίου του άνθρακα. Θα ακούσουμε την παρουσίαση μιας μελέτης ε, που την διαχειρίστηκε το Τμήμα Πολιτικής ή Τμήμα Πολιτικών μάλλον. Ένας από τους συντάκτες της έκθεσης θα μας κάνει και τη σχετική παρουσίαση. Ο ποιος έπρεπε να ρωτήσω γιατί δεν είμαι σίγουρος για την προφορά του ονόματος του καλεσμένου μας. Λέγεται κουν Rademakers και είναι διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας Trinomics. Πριν γίνει σύμβουλος, εργάστηκε ως επίκουρος καθηγητής στο Πανεπιστήμιο των Βρυξελών. Επίσης, ήταν υπεύθυνο ε, για θέματα οικονομικών ενέργειας και κλιματικών αλλαγών στο υπουργό, στο Φλαμανδό Υπουργό Οικονομικών, στο γραφείο του Φλαμανδού Υπουργού Οικονομικών. Και τα τελευταία δέκα χρόνια ο κύριος Ράντε Μάκερς ε, ηγήθηκε σχεδίων για θέματα ενεργειακής πολιτικής και συναφή ζητήματα ε, και κυρίως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο δεύτερος από τους δύο συντάκτες της έκθεσης είναι ο κύριος Λουκ Βανούφελ. Και οι δύο ε, συντάκτες εξέτασαν το πώς η σύζευξη των τομέων μπορεί να αυξήσει την, ε, ε, την καλύτερη ενσωμάτωση και την καλύτερη ολοκλήρωση των δικτύων τελικής χρήσης και παροχής και την αύξηση της, αποφασ... αποτελεσματικότητας και της ελαστικότητας των ενεργειακών συστημάτων καθώς και της αξιοπιστίας και της επάρκειάς τους. Επίσης, η σύνδευξη των τομέων μπορεί να μειώσει το κόστος τη ε, απαλλαγή μα από τις ε, εκπομπές του εξουδίου του άνθρακα. Πολύ ενδιαφέρον θέμα. Θα ήθελα λοιπόν να σας δώσω το λόγο για να μα κάνετε την παρουσία σα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα μια σύντομη εισαγωγή ε, στην εταιρεία μας, στην Trinomics. Κυρίως ε, παρακολουθούμε ενεργειακά σχέδια και σχέδια χρηματοδότηση ενέργεια υπό την αιγύδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και βοηθούμε τη Γενική Διεύθυνση ε, Κλίματος για να αποτρέψουμε τις διαρροές ε, άνθρακα και ασχολούμαστε κυρίως ε, με κλιματικά και περιβαλλοντικά ζητήματα. Το θέμα στη σημερινή ακρόαση είναι πώς η σύζευξη των τομέων μπορεί να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και τη σταθερότητα του δικτύου και να ε, ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα. Καταρχήν, τι η συζεύξη των κλάδων. Η βασική πρωτοβουλία προήλθε από τη Γερμανία και αφορούσε κυρίως την ηλεκτροδότηση των τομέων τελικής χρήσης. Δηλαδή, προσπαθούμε να διαπιστώσουμε και να ε, καταφέρουμε να καλύψουμε τις ανάγκες των διαφόρων ε, τομέων και να καλύψουμε όλες τις ανάγκες σε ενέργεια, στα κτίρια, στις μεταφορές και στη βιομηχανία. Επίσης, το θέμα της σύζευξης τομέων μπορούμε να το δούμε υπό ευρύτερη προπτική στα ενεργειακά συστήματα και την ολοκλήρωσή τους. Βλέπετε λοιπόν ότι έχουμε δύο διαφορετικούς ορισμούς, για να μην πω πολύ περισσότερους ορισμούς για τη σύζευξη των τομέων, αλλά εμείς τους εξετάζουμε ε, κυρίως ε, υπό το πρίσμα της ε, σύζευξης τομέων τελικής χρήσης και την σύζευξη μεταξύ των φορέων. Έχουμε την ηλεκτροδότηση της ζήτησης, ενώ ισχύουμε την διάδραση μεταξύ της παροχής και της τελικής χρήσης και μετά έχουμε μια ολοκληρωμένη χρήση ενέργειας υποδομών και φορέων και ιδιαίτερα της ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, μας ενδιαφέρει το θέμα της αποθήκευσης, αλλά εξετάζουμε και τρόπους μεταφοράς και αποθήκευσης ενέργειας. Αυτά είναι τα βασικά σημεία της έκθεσης, οι βασικοί άξονες της έκθεσης. Και αυτό που σας εξήγησα το βλέπουμε και στην διαφάνεια που βλέπετε. Εξετάζουμε πρώτα αφενός την προσφορά, την παροχή της ενέργειας, μετά έχουμε τους φορείς ενέργειας, ε, ή, ή τη μεταφορά ή την αποθήκευση και έχουμε και την τελική χρήση, τους κλάδους της τελικής χρήσης. Προσπαθούμε λοιπόν να βελτιστοποιήσουμε στο μέλλον και όλες τις στρατηγικές μας ε, εν ώψη το 2030-2050 και μάλιστα χάρη στη σύζευξη με ε, αποτελεσματικό τρόπο και με τρόπο που να πιάνουν το από τα κονδύλια που έχουμε. Ο κύριος Λουκνεφέλ, σε αυτή τη διαφάνεια εξηγούμε πόσο σημαντική έχει γίνει η σύζευξη των τομέων, ιδιαίτερα στη στρατηγική και για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Διαπιστώνουμε ότι ήδη το 2017 σε κάποια κράτη-μέλη η ΑΠΕ και οι ικανότητε ΑΠΕ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας είναι μεγαλύτερη από το μέγιστο φορτίο, τη μέγιστη κατανάλωση δηλαδή. Κάτι που σημαίνει ότι κάποιες ώρες της ημέρα υπάρχει ανάγκη αποθήκευσης ενέργειας που είναι πλεονασματική ή της μετατροπής της ηλεκτρικής ενέργειας σε άλλους φόρου ενέργεια, ώστε να μπορεί να μεταφερθεί ή να αποθηκευτεί ή να χρησιμοποιηθεί για άλλες τελικές χρήσεις. Με άλλα λόγια, Χρειαζόμαστε στρατηγικές και τεχνολογίες προκειμένου να αξιοποιήσουμε το πλεόνασμα ενέργειας που έχουμε και δεν το χρειαζόμαστε. Και αυτές οι στρατηγικές ε, θα πρέπει να αφορούν πιο ελαστική παραγωγή ενέργειας, ε, να ανταποκρίνονται στη ζήτηση, στην, στα, στις ανάγκες αποθήκευσης και στη μετατροπή ενέργειας σε αέριο καύσιμο. Mm. Μετατροπή ηλεκτρισμού σε αέριο Τώρα, εδώ έχουμε τον αντίκτυπο της πλεονασματικής παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στις αγορές. Διαπιστώνουμε ότι πέρυσι, για παράδειγμα, περίπου, 10, περίπου 70 ώρες είχαμε αρνητικέ τιμές στην αγορά, σε κάποιες αγορές τουλάχιστον. Όχι σε όλες τις περιφέρειες, σε όλα τα κράτη-μέλη. Ε, αλλά σε κάποιες χώρες όπου η δίσδυση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας ήταν υψηλή, διαπιστώσαμε ότι είχε πρόβλημα με τις αρνητικές τιμές λόγω πλεονασματικής πλεονάζουσας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Θεωρούμε ότι αν οι τιμές είναι αρνητικές ή χαμηλότερες από ένα ε, ελάχιστο κατόφλι, 20 ευρώ την κιλοβατόρα, θα είχε νόημα από οικονομική άποψη να μετατρέψουμε αυτή την πλεονασματική ηλεκτρική ενέργεια σε άλλους φορείς ενέργειας, για παράδειγμα ανανεώσιμο αέριο. Τώρα άλλο θέμα που συνηγορεί υπέρ της προώθησης της σύζευξης τομέων που τη θεωρούμε καλή στρατηγική. Σχετίζεται με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με το αέριο. Από τη μία πλευρά και από την άλλη πλευρά αφορά τα χαρακτηριστικά της τελικής χρήσης. Στις μεταφορές, για παράδειγμα, τα ΙΧ τα επιβατικά οχήματα μπορούν να αντικατασταθούν από ηλεκτρικά οχήματα, αλλά για τις μεταφορές σε εμπαρευματικές, με την αυτιλία ή την αεροπορία, αλλά και για τις ε, οδικές μεταφορές ε, μεγάλων αποστάσεων, εκεί η ηλεκτροδότηση, οι ηλεκτρικές μεταφορές δεν είναι κατάλληλη λύση. Το βιομεθάνιο ίσως ή το υδρογόνο θα μπορούσαν εκεί να είναι πιο κατάλληλη τρόποι, καταλληλότερες λύσεις. Επίσης, έχουμε κάποιες ειδικέ τελικές χρήσεις στη βιομηχανία που επίσης δεν μπορούν να καλυφθούν από ηλεκτρική ενέργεια. Για παράδειγμα, θέρμανση σε πολύ ψηλέ θερμοκρασίε, αλλά και χρήση υδρογονανθράκων σε κάποιε βιομηχανίε, όπω τη χημική βιομηχανία, στα λοιπάσματα ή στα χημικά προϊόντα. Αυτό είναι ο λόγο λοιπόν για τον οποίο θα μπορούσαμε να ε, θεωρήσουμε τη σύζευξη τομέων ως πολύ καλή λύση. Και δεύτερο επιχείρημα προς αυτήν την κατεύθυνση είναι ε, ένα επιχείρημα συναφές με τα χαρακτηριστικά. Βλέπετε στις γραφικές παραστάσεις ότι το ελάχιστο ε, ως προς το μέγιστο φορτίο ηλεκτρικής ενέργειας σε σχέση με το αντίστοιχο φορτίο ελάχιστο και μέγιστο του αερίου είναι πολύ διαφορετικά. Το μέγιστο φορτίο αερίου είναι εφταπλάσιο από το ελάχιστο φορτίο σε ημερήσια βάση από, την, από τον ηλεκτρισμό. Και βλέπουμε τα στοιχεία μηνιαίος, αλλά για να έχουμε μια ιδέα των περιορισμών των ικανοτήτων θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το ημερήσιο φορτίο για το αέριο αφενός, που είναι ένα προς 7, 7 πλάσιο δηλαδή, και το ωραίο φορτίο για, τον ηλεκτρισμό. Αυτό είναι, αυτά είναι πολύ βασικά στοιχεία που προσδιορίζουν τους περιορισμούς στην ικανότητα. Και τα ωραία όρια εκεί για τον ηλεκτρισμό τουλάχιστον είναι 2 προς 1. Δηλαδή το μέγιστο φορτίο στην ηλεκτρική ενέργεια είναι διπλάσιο από το... Ε, το μέγιστο φορτίο είναι ε, διπλάσιο από το μέγιστο φορτίο στον ηλεκτρισμό. Οπότε εκεί που θα πρέπει η κατανάλωση αερίου να αντικατασταθεί από ηλεκτρική ενέργεια θα πρέπει να έχουμε καλές υποδομές, ε, μεταφορές, αποθήκευση που θα είναι τετραπλάσεις ε, από, την, ε, ισχύους, από τις ισχύουσες ικανότητες των υποδομών. Αυτός ο τετραπλασιασμός των εκατοτήτων είναι υπερβολικά δαπανηρός και οικονομικά ανέφικτος. Και γι' αυτό λέμε ότι θα πρέπει να, να κάνουμε μια σύζευξη, ένα συνδυασμό των τομέων της παραγωγής και της μεταφοράς που θα των φορέων μάλλον ενέργειας και αυτό θα ήταν καλή λύση για να αποφύγουμε την αντικατάσταση. Στη διαφάνεια αυτή επικεντρωνόμαστε σε κάποιες τεχνολογίες, τις ε, βασικές τεχνολογίες και τις βασικές τεχνολογικές επιλογές που έχουμε για να καταφέρουμε να υλοποιήσουμε τη μετάβαση σε μια ενεργειακή κατάσταση που δεν θα χρησιμοποιεί, θα παράγει διοξίδιο του άνθρακα. Έχουμε αφενός την ηλεκτροδότηση, ε, του ε, τομέα μεταφορών αλλά και των κατοικιών. Εκεί δύο είναι ηγετικέ τεχνολογίες, τα ηλεκτρικά οχήματα και οι αντιλίε θερμότητας και η σύζευξη των τομέων ηλεκτρισμού και αερίου. Εκεί έχουμε τα δύο πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα που είναι το power to gas και power to liquids, μετατροπή ηλεκτρική ενέργειας σε υγρό ή αεροκαύσιμο και το CCS που είναι αποθήκευση και μεταφο... Ε, δέσμευση, χρήση και αποθήκευση του άνθρακα. Όχι μόνο στις βιομηχανικές διαδικασίες ή στην παραγωγή ενέργειας, αλλά με ολοκληρωμένο τρόπο που παίζει το ρόλο του και στη σύζευξη των τομέων. Όπως είπα λοιπόν, όταν έχουμε πλεονάζουσα ηλεκτρική ενέργεια και αρνητικές τιμές, θα πρέπει να μπορούμε να τη μετατρέψουμε σε υδρογόνο αυτή την ηλεκτρική ενέργεια και να την διοχετεύσουμε άμεσα στο δίκτυο αερίου ή να την ε, αποθηκεύσουμε τοπικά ή μπορούμε να την μετατρέψουμε σε συνθετικό αέριο που έχει και το πλεονέκτημα ότι έχει ακριβώς τα ίδια χαρακτηριστικά με το φυσικό αέριο που χρησιμοποιούμε άρα δεν θα επηρεάσει καθόλου ούτε τις υποδομές ούτε τις εφαρμογές τελικής χρήσης αλλά το μειονέκτημα είναι το υψηλότερο κόστος του συνθετικού αερίου σε σχέση με το φυσικό. Οπότε θα πρέπει να βρούμε ε, πώς θα αντισταθμίσουμε το κόστος, λαμβάνοντας υπόψη και τα, τον περιβαλλοντικό αντίκτυπο και τον αντίκτυπο στους χρήστες. Επίσης, η ηλεκτρική ενέργεια μπορεί να μετατραπεί σε υγρά καύσιμα, μεθανόλη για παράδειγμα, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στις οδικές μεταφορές, στις μεταφορές γενικώς. Αυτά είναι μερικά παραδείγματα τεχνολογιών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στα πλαίσια αυτού του συνδυασμού των τομέων, τη σύζευξη των τομέων και μάλιστα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στους διάφορους τομείς που αναφέρονται εδώ στα δεξιά, στο δεξιό τμήμα της διαφάνειας. Σε αυτό το πλαίσιο λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να επικεντρωθούμε στον δυνητικό ρόλο του ανανεώσιμου αερίου στην στο μέλλον της προσφοράς ενέργειας, παροχής ενέργειας. Έχει τεράστια πλεονεκτήματα και ως προς την ελαστικότητα, ε, ως εφεδρεία για την ηλεκτρική ενέργεια. Επίσης και για την αποθήκευση έχει πλεονεκτήματα. Το δυναμικό αποθήκευσης του αερίου είναι τεράστιο. Το ισχύον δυναμικό αποθήκευση σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι το 1 τρίτο της ε, τρέχουσας κατανάλωσης. Βλέπετε τεράστιο δυναμικό αποθήκευσης που υπάρχει και που θα εξασφαλίσει ελαστικότητα των ενεργειακών συστημάτων. 1100 τεραβατ, την ώρα. Ένα τρίτο δηλαδή της ισχύουσας ε, ηλεκτρικής ικανότητας. Ενώ το δυναμικό αποθήκευση ηλεκτρικής ενέργειας είναι πολύ περιορισμένο, μόνο 600 ΜΒ σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μεγάλη διαφορά. Και θα πρέπει το θέμα της ικανότητας αποθήκευσης στο μέλλον να τη, βάλουμε, να τη λάβουμε υπόψη για την παροχή ενέργειας. Για να αποφύγουμε τη δημιουργία νέα ικανότητα για την αποθήκευση ηλεκτρισμού που δεν συμφέρει σε σχέση με την αποθήκευση του αέριου. Οπότε φαντάζεστε ότι στο πλαίσιο αυτό η σύζευξη ηλεκτρισμού και αερίου ε, θα μπορούσαμε στο μέλλον, στα, την επόμενη 20 ετία, στα επόμενα 20-30 χρόνια, ε, συνδυασμό ανεμογεννητρίων με αποθήκευση υδρογόνου και να μεταφέρουμε την ενέργεια με το καύσιμο υδρογόνου προς τελικούς χρήστες ως αέριο. Γιατί ένα προς δύο είναι η τιμή της μεταφοράς στο αέριο σχέση με τον ηλεκτρισμό. Άλλο πολύ σημαντικό σημείο πάλι στο θέμα της σύζυγης των τομέων είναι αυτή η ηλεκτροδότηση, η χρήση ηλεκτρικής ενέργειας. Και εδώ έχουμε δύο παραδείγματα που το αποδεικνύουν. Καταρχήν, τα ηλεκτρικά οχήματα. Αν αντικαταστήσουμε τα, τους κινητήρες των οχημάτων με ηλεκτρικά οχήματα, θα αυξηθεί κατά 140 περίπου το 100 και παραπάνω ίσως η αποτελεσματικότητά σας. Αυτό είναι αρκετά πιστικό επιχείρημα. Βέβαια θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και τον οικονομικό αντίκτυπο. Αυτό είναι ένας αντίκτυπος που σας δίνει η αποτελεσματικότητα, που θα είναι πάνω από 140, 144%. Θα έχουμε μικρότερη κατανάλωση ενέργειας, λιγότερα αέρια του θερμοκηπίου και κάτι άλλο πολύ σημαντικό, θα έχουμε και λιγότερη εκπομπή υπογόνων ουσιών πέραν του διοξίδιου του άνθρακα. Αυτό είναι ένα παράδειγμα. Επίσης, ε, αντιλίες θερμότητας. Αν αντικαταστήσουμε τους ε, καυστήρες συμπυκνωμένου αερίου που έχουν υψηλή αποτελεσματικότητα, αν τους αντικαταστήσουμε παρόλα αυτά από ηλεκτρικές αντιλίες θερμότητας, θα έχουμε τριπλάσια εξοικονόμηση αποτελεσματικότητας τριπλάσια αποτελεσματικότητα. Ο συντελεστής απόδοσης ε, των ε, θερμοαντλιών είναι 300%. σε σχέση με την αποτελεσματικότητα της ηλεκτρικής ε, ενέργειας που είναι 100%. Είναι τριπλάσια η αποτελεσματικότητα των θερμοαντλειών. Είχατε ένα τέταρτο, το εξαντλήσατε, παρακαλώ να ολοκληρώσετε ίσως ε, κάποια συμπεράσματα για το τέλος. Πολύ γρήγορα τότε να περάσω στις υπόλοιπες διαφάνειες. Εδώ δίνουμε έμφαση στην ευελιξία λοιπόν. Όμως νομίζω πως ε, είναι προφανές ότι η αποθήκευση ανάλογα με την ε, ζήτηση λοιπά είναι τεχνολογίες λίγο πολύ γνωστές. Και είναι γνωστό ότι συνεισφέρουν σε αυτήν την αναγκαία ευελιξία στον ε, τομέα της ε, ηλεκτροδότησης, αλλά και αυξάνουν την ε, χρήση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Νομίζω πως είναι αυτονόητο όλα αυτά και δεν χρειάζεται να τα εξηγήσουμε περαιτέρω. Όμως, είναι σημαντικό να τονίσουμε τον αντίκτυπο της σύζευξης τομέων στο συνολικό κόστος. Ήδη αναφέρθηκα στο ότι αν χρησιμοποιήσουμε αυτήν την σύζευξη, τότε θα υπάρξει ανάγκη για νέες υποδομές, καλύτερες υποδομές ε, παραγωγής ενέργειας και δικτύων, ε, επέκταση των ε, υφιστάμενων δικτύων. Εδώ βλέπετε τα αποτελέσματα μιας μελέτης η οποία έγινε στη Γερμανία, η οποία συμπεραίνει ότι ακόμα και σε περίπτωση που ο στόχος είναι 95% λιγότερες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, το συνολικό κόστος είναι χαμηλότερο από τα άλλα σενάρια, όπου δηλαδή ο στόχος μείωσης εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου είναι μόνο 80%. αναφερόμενοι στην, ε, στον εξηλεκτρισμό της χρήσης καυσίμων. Εδώ βλέπετε λοιπόν τον αντίκτυπο και τις ε, θετικές επιπτώσεις της σύζευξης τομέων. Αυτή η μελέτη στηρίζεται και από άλλες μελέτες, ε, από μια μελέτη της ε, Euroelectric, της Ένωσης Εκπροσώπων της Βιομηχανίας Ηλεκτρισμού και Ηλεκτροδότησης και νομίζω πως το αποτέλεσμα δείχνει πως αυτή είναι η καταλληλότερη επιλογή. Και τώρα θα περάσουμε στους φραγμούς και τα εμπόδια τα οποία πρέπει να αντιμετωπιστούν νομοθετικά τα κυριότερα εμπόδια αυτή τη στιγμή έχουν να κάνουν με το κόστος και τις επιδόσεις που φυσικά συνδέονται και αφορούν την έλλειψη υποδομών, τεχνικών υποδομών και οικονομικών. Μετά, πολιτική. Εδώ υπάρχουν εμπόδια στον σχεδιασμό που θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν νομοθετικά. Η δική μας πρόταση λοιπόν είναι να εστιάσουμε σε αυτό το σκέλος. Και τέλος βλέπουμε τις ε, συστάσεις ε, σε υψηλό επίπεδο. Εδώ βλέπετε μία σύνοψη των ε, συστάσεων. Φυσικά πρώτη σύσταση είναι να αντιμετωπιστούν τα εμπόδια και οι προκλήσεις. Τελευταία διαφάνεια είναι αυτή που θα σας δείξω. Η πρώτη σύσταση πολιτικής λοιπόν αφορά την ανάγκη για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση στο σχεδιασμό αλλά και στο λειτουργικό στάδιο που θα περιλαμβάνει αξιολόγηση των επενδύσεων ε, με βάση τις εναλλακτικέ λύσεις που υπάρχουν. Για παράδειγμα, αν μια επένδυση ε, στο τομέα του ηλεκτρισμού είναι υπό εξέταση, θα πρέπει να ε, εξεταστούν και άλλες εναλλακτικέ λύσεις που θα χρησιμοποιούν τις ήδη υπάρχουσες υποδομές αερίου, για παράδειγμα. Όλες οι επενδύσεις θα πρέπει να είναι θωρακισμένες ως προς τις μελλοντικές προκλήσεις, δηλαδή τι εννοούμε με αυτό, ότι οι επενδύσεις θα πρέπει να είναι κατάλληλες και για μελλοντικές χρήσεις ενέργειας, για αποθήκευση δρογόνου για παράδειγμα. Μετά, παρατηρούμε πως υπάρχει ανάγκη για αυξημένη χρήση των ε, έξυπνων, της έξυπνης τεχνολογίας, έτσι ώστε να διευκολυνθεί αυτή η σύζευξη τομέων. Θα πρέπει να ενισχυθεί η χρήση των νέων τεχνολογιών, ιδιαίτερα του υδρογόνου. Και μετά αναφέρονται ορισμένε συστάσεις θέματα marketing. Αναφερόμαστε στη νέα δέσμη μέτρων για τον ε, σχεδιασμό διάθεση στην αγορά και επίσης τονίζουμε πως υπάρχει ανάγκη για περισσότερη έρευνα και ανάπτυξη με έμφαση στις καινοτομές τεχνολογίες, ιδιαίτερα τις τεχνολογίες υδρογόνου, έτσι ώστε να μειωθεί το κόστος και να γίνει πιο εύκολη η ανάπτυξη αυτής της τεχνολογίας σε, ε, μεγάλο, ε, μεγάλη έκταση. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίασή σας σχετικά με το κόστος της ενεργειακής μετάβασης. Τώρα, αγαπητοί συνάδελφοι, έχετε ερωτήσεις ή σχόλια. Ο κύριος Κόβιτσέκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πρόεδρε. Θα ξέρετε ότι είμαι μηχανικός. Λοιπόν, είχα τη θεωρία των καυστήρων, των υψικαμίνων, στη θέση που έγραψα. Λοιπόν, θα πρέπει να εξετάσουμε βήμα-βήμα αυτά που μας παρουσιάσατε, λέξη-λέξη κανονικά και θα χρειαζόταν δύο-τρεις ώρες. Διότι δεν είναι πολύ αναλυτικές κάποιες δηλώσεις σας. Όταν τα βλέπει ένας μηχανικός, οι δικαιοκριμένοι συνάδελφοι που δεν είναι μηχανικοί θα μπορούν να πούν ότι αυτά που μας είπατε είναι αρκετά. Πρώτα απ' όλα, για πρώτη φορά είναι υπέροχο να ακούς κάποιον στην ομιλία του να, να λέει επανειλημμένα τη λέξη υδρογόνο. Για πρώτη φορά στην Επιτροπή μας. Δεύτερον, 1% της ενέργειας πρέπει να αποθηκεύεται σε υδρογόνο. Μέχρι το 2020. Είναι απόφαση ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που ελήφθη εδώ και κάποια χρόνια. Ελπίζουμε να ισχύει. Τρίτον, μεταφορά σε μεγάλες αποστάσεις. Συμφωνώ, υπάρχουν απώλειες. Στο ρεύμα υψηλή τάσεω, υψηλότερη απώλεια από ό,τι σωλήνων Η απώλεια ενέργεια είναι μεγαλύτερη. Κάτι δεν είναι ξεκάθαρο. Α πούμε, χρησιμοποιείται έναν αγωγό για μεθάνιο. Ανεξάρτητα είναι βιομεθάνιο ή φυσικό αέριο. Λόγω προσθήκων. που κάποια άλλα συστατικά είναι στο φυσικό αέριο και όχι στο βιομεθάνιο, άλλη σύνθεση το ένα, άλλη σύνθεση το άλλο. Αλλά δεν υπάρχει πρόβλημα. Το υδρογόνο χρειάζεται άλλες αντλίες. Πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί διότι uh, uh, έχει ιδιαιτερότητες το υδρογόνο. Στη Γερμανία μπορεί να προσθεθεί μέχρι 7% υδρογόνο στο φυσικό αέριο. Εγώ όμως, σαν κάποιος που διόρθωνε και παρήγαγε για αυτούς τους υψηκαμίνους, ξέρουμε ότι έχει πολύ μικρή και ισχυρή φλόγα, ενώ το μεθάνιο δεν είναι τόσο επιθετικό το ΣΥΠΗΝ. Το ένα παράγει μια φλόγα που είναι πολύ, αν θέλουμε να έχουμε μια φλόγα που να είναι μακριά και πιο λαμπρή το μεθάνιο είναι καλύτερο. Και είναι και το θέμα και... είναι και η χρήση, αν θέλουμε να λιώνουμε γυαλί φερρυπίν ή παραγωγή κεραμικών. Αντίθετα, το φυσικό αέριο είναι καλό, το μεθάνιο. Το υδρογόνο έχει διαφορετικές ιδιότητες και τιμές όταν χρησιμοποιείται στην τεχνολογία. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε πλοία, αεροσκάφη, αερομεταφορές κλπ διάφορα παραδείγματα. Μεταφορά διαπλοίων. Στα πλοία χρησιμοποιείται η ολική ενέργεια. Έχουμε ελιοσυσσωρευτές κλπ. Όλα αυτά θα είναι πολύ σημαντικά για το μέλλον. Η ολική ενέργεια και οι συσσωρευτές. Έχουμε κάποια αεροσκάφη, πολύ ελαφρά, που χρησιμοποιούν ηλεκτρική ενέργεια από, τις, από ηλιοσυσσωρευτές και μπορούν να ταξιδέψουν σε όλο τον κόσμο αυτά τα μικρά αεροσκάφη. Ίσως στο μέλλον μπορούμε να παράγουμε από αυτές τις ηλιακές κυψέλες καλύτερη ενέργεια. Έχουμε καλύτερη αποδοτικότητα και μπορεί να λειτουργήσει αυτή η λύση. Αλλά για την ώρα έχετε δίκιο. Λοιπόν, η ολοκληρωμένη προσέγγιση. Ένα παράδειγμα στη Βιέννη χρησιμοποιείται. Ε, μια συνοικία της πόλης, κοντά στο διεθνές αεροδρόμιο, έχει σχεδιαστεί με αποθήκευση ενέργειας σε ζεστό νερό. Λαμπρό παράδειγμα για μικρές πόλεις, μέχρι 2 εκατομμύρια κατοίκους. Που μπορεί να γίνει αυτό και στην Ευρώπη. Σας ευχαριστώ πολύ. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρέμβασή σας, όμως θα χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο και να μπούμε σε βάθος. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, ευχαριστώ συνάδελφοι για τα σχόλιά σα. Για μένα υπάρχει κάτι πολύ ενδιαφέρον. Αναφερθήκατε σε δύο τομείς. Τελική χρήση ενέργεια και εφοδιασμό. Ο σχετικό τομέα Και άλλος σημαντικός τομέα. Ο ψηφιακή τομής. χωρίς ευφύς λύσεις δεν μπορούμε να προχωρήσουμε. Αυτό είναι απλώς ένα σχόλιο. Ο κ. Φρόιντ, ευχαριστώ. Ζητώ συγγνώμη που άργησα λίγο. Δεν άκουσα όλη την παρέμβαση. Αναφερθήκατε στο υδρογόνο. Το ανέφερε και ο συνάδελφος. Πολύ ενδιαφέρον θέμα. Όλοι γνωρίζουμε ότι επί του παρόντος υφίσταται τεχνολογία, όπου εκεί το υδρογόνο παίζει πολύ σημαντικό ρόλο όσον αφορά την μετατροπή της ενέργειας. Οι κυψέλες καυσίμων εξαρτώνται από το υδρογόνο. Αυτό διευκολύνει μεταφορά ε, απόσταση να καλύπτεται πάνω από 300 χιλιόμετρα. Αυτή είναι η απόσταση που καλύπτεται από τις μπαταρίες. Ξέρω ότι από εκεί που προέρχομαι μπορεί να αγοράσει κανείς αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν κυψέλες ενέργειας με υδρογόνο. Δύο διαφορετικές μάρκες μπορεί να αγοράσει. Αλλά σε όλη την Αυστρία υπάρχουν μόνο τρει σταθμοί όπου μπορεί να πα και να γεμίσει το ρεζερβουάρ με υδρογόνο. Δεν ξέρω αν αυτό είναι μια παράκαμψη για το μέλλον των μεταφορών, δηλαδή πάνε πρώτα από την μπαταρία, μετά στις κυψέλες καυσίμων και μετά κάτι άλλο θα προκύψει. Ή και εσεί θεωρείτε ότι το υδρογόνο και αυτές οι κυψελίδε καυσίμων θα μας δώσουν το καλύτερο σύστημα για τις μεταφορές στην Ευρώπη και στον υπόλοιπο κόσμο. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Έχουμε μέλη της κοινότητας του Σαν Κάντσιαν από την Καρινθία της Αυστρίας. Ήρθαν εδώ να μας ε, επισκεφτούν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καλώς ήρθατε, δεν βλέπω που κάθεστε. Καλώς μας ήρθατε, μπράβο σας. Τους προσκάλεσε ο συνάδελφος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, ο κύριος Όγγεν Φρόιντ. Θερμά χειροκροτήματα σε όλους κύριος Φρόιντ εκπροσωπεί τους ψηφοφόρους, τους συμπολίτες του και χαίρομαι που οι συμπολίτες του είναι εδώ για να ακούσουν τις συζητήσεις μας. Τώρα θα δώσω το λόγο στους καλεσμένους μας, στους συντάκτες της εργασίας αυτής, ε, για να μας κάνουν σύντομα σχόλια μετά τις ερωτήσεις που ακούσαμε από την Ομιγύρη. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ και για τα σχόλια και για τις ερωτήσεις σας. Έχετε απόλυτο δίκιο. Κατά, μάλλον ο τρόπος με τον οποίο παρουσιάσαμε τη λύση του υδρογόνου παρά ήταν αισιόδοξο, ήταν υπεραισιόδοξο ο τρόπο και σίγουρα δεν πρόκειται να γίνει πραγματικότητα το 2020 ούτε καν πριν το 2030. Πάντως θεωρούμε ότι είναι ρεαλιστική η επιλογή το υδρογόνο μετά το 2030. Βέβαια ακόμη έχουμε πολλά εμπόδια και φραγμούς, εκτός από το κόστος, που είναι φυσικά κρίσιμο στοιχείο, το, η δυνατότητα αναβάθμιση των, των υποδομών, των εγκαταστάσεων, ε, το θέμα των ικανοτήτων. Υπάρχουν πολλές εκκρεμότητες που θα πρέπει να διευθετηθούν μέχρι ότου γίνει το υδρογόνο κατάλληλη λύση για το μελλοντικό μας ενεργειακό μείγμα και τα ενεργειακά μας συστήματα. Αναφερθήκατε σε κάποια προβλήματα στις, ε, στο θέμα της πίεσης, της ιδιαιτερότητας του υδρογόνου σε σχέση με το βιομεθάνιο και το φυσικό αέριο. Ε, και αυτό είναι ο λόγος ε, για τον οποίο εξετάζουμε διάφορε επιλογές. Μία επιλογή θα μπορούσε να είναι συστήματα διανομής για το υδρογόνο, καθώς και συγκεκριμένε ε, συσκευέ τελικής χρήσης. Και άλλο ήταν να μετατρέψουμε το υδρογόνο σε συνθετικό μεθάνιο, που έχει τα ίδια χαρακτηριστικά ακριβώς, αλλά και υπάρχει το κόστος που είναι απαγορευτικό. Και τρίτο θέμα είναι να ε, μεταφέρουμε το υδρογόνο στο, ε, στο δίκτυο του αερίου. Εκεί όμως έχουμε διαφορετικά χαρακτηριστικά των υποδομών ε, της διανομής και της μεταφοράς και ως προς συσκευές τελικής χρήσης. Το πρόβλημα όμως είναι και οικονομικό, γιατί αν μεταφέρουμε το υδρογόνο στο δίκτυο αερίου, δεν μπορούμε να ε, κάνουμε απολογισμό της τελική αξίας του προϊόντος σε σχέση με το... και να συγκρίνουμε τις αξίες των δύο προϊόντων, αφού θα έχει μπει και το υδρογόνο στο δίκτυο του αερίου. Αυτά τα θέματα λοιπόν θα πρέπει να το δούμε, όπως και το ζήτημα των προσμίξεων που είπατε προηγουμένως. Άλλο θέμα που αφορά το ρόλο στο μέλλον των κυψελών καυσίμου. Θεωρούμε ότι οι κυψέλες καυσίμου εδώ και 10-20 χρόνια ε, κρίθηκαν ως ε, κατάλληλη λύση για τις κατοικίες, για τη θέρμανση κατοικιών, αλλά πλέον δεν θεωρούνται ως βιώσιμη λύση η πολλά υποσχόμενη ελπιδοφόρα λύση για την Ευρώπη, ενώ σε άλλες υπήρους ε, είναι επιτυχημένη επιλογή. Είναι κάπως περίεργο που και παράδοξο που εμείς στραφήκαμε σε άλλες τεχνολογίες και σε άλλες λύσεις και εγκαταλείψαμε πια το θέμα των κεψελών καυσίμου. Σε ό,τι αφορά τις κεψέλες καυσίμου για το τομέα των μεταφορών, συμφωνώ απόλυτα ότι δεν έχουμε αφενός αρκετά οχήματα. Η Hyundai, αν δεν κάνω λάθος, έχει θέση κυκλοφορία κάποια οχήματα που χρησιμοποιούν κυψέλες καυσίμου, αλλά λίγα, γιατί δεν υπάρχουν υποδομές. Θεωρούμε ότι αυτή η λύση είναι πιο κατάλληλη για εμπορευματικές μεταφορές, για φορτικά και ενταλίκες περισσότερο παρά για επιβατικά οχήματα ή γιοταχή. Σας ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε θερμά. Ή θέλετε να προσθέσετε και εσείς κάτι. Να πω κάποια γενικά σχόλια για τη μελέτη μας. Πρόκειται για μία μελέτη που κάνει μια γενική επισκόπηση του ζητήματος της σύζευξης τομέων περιγράφει την κατάσταση και κάποιες δυνατότητες. Είχαμε και περιορισμό ε, μεγέθους. Δεν μπορούσαμε να ξεπεράσουμε τις 50 σελίδες, γι' αυτό και δεν ήμασταν διεξοδίκοι σε όλα τα σημεία. Ίσως στην... η επόμενη επιτροπή, στο νέο κοινοβούλιο ε, και η νέα επιτροπή θα μπορούσαν να εγκύψουν στο θέμα αυτό, γιατί έχουμε και τα εθνικά σχέδια ενέργειας και κλίματος. Ίσως Εκεί θα μπορούσε να γίνει μια καλύτερη επισκόπηση για το τι σκοπεύουν τα κράτη-μέλη να κάνουν στα θέματα αυτά και τι είναι εφικτό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο για να δούμε πού υπάρχουν κενά, δυναμίες αλλά και τι συνέργειες μπορούν να προκύψουν από τα εθνικά σχέδια ενέργειας και περιβάλλοντος και μετά να δούμε και τις επενδύσεις. Πάντως αυτό λείπει προς το παρόν. Να δούμε πώς θα διαμορφωθούν τα εθνικά σχέδια και μετά να κάνουμε ένα βήμα και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ λοιπόν για την παρουσίασή σας αλλά και την εξαιρετική σας ε, έκθεση. Μπράβο σας λοιπόν, πολύ καλή δουλειά, πολύ χρήσιμη για όλους μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητοί φίλοι, πρωτού περάσουμε στις ψηφοφορίες τη 4, έχουμε άλλο ένα θέμα να συζητήσουμε για την ενεργειακή επισήμανση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μας παρουσιάσει μια δέσμη κατεξουσιοδότηση πράξεων για πέντε ομάδες προϊόντων προτεραιότητας πλυντήρια πιάτων, πλυντήρια ρούχων, ψυγεία, φωτισμό και τηλεοράσεις. Η παρουσίαση θα γίνει από τον Hans Van Skin, Διευθυντή στην Γενική Διεύθυνση Ενέργειας. Αγαπητέ για αυτό το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Μπούσε, Καλησπέρα σε όλους. Ε, δεν έχουμε πολύ χρόνο από το καταλαβαίνω, οπότε θα προσπαθήσω να είμαι γρήγορος. Είναι όμω ένα σημαντικό θέμα το οποίο πρέπει να συζητήσουμε. Θα σας παρουσιάσω λοιπόν τη, αυτά που ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 4 Μαρτίου σχετικά με την νέα επισήμανση ηλεκτρικών συσκευών. Είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της ε, Ενεργειακής Ένωσης στοχεύει μεταξύ άλλων να ε, δώσει την ε, δύναμη πάλι στους καταναλωτές. Η ενέργεια είναι ένας τρόπος να γίνει αυτό, να χειραφετηθούν οι καταναλωτές, ε, διότι από τη μία η, ενέργεια, η ξεκάθαρη ενεργειακή σήμανση θα δώσει στους καταναλωτές τη δυνατότητα να συγκρίνουν πληροφορίες και προϊόντα, να συγκρίνουν τις ενεργειακές επιδόσεις λοιπόν των προϊόντων αυτών, έτσι ώστε όταν αγοράζουν ένα νέο ψυγείο, ένα νέο πλυντήριο, να ε, ξέρουν τι αγοράζουν. Το σημαντικό είναι ότι αυτή η επισήμανση έχει βελτιώσει τον ε, ανταγωνισμό μεταξύ ε, επιχειρήσεων έτσι ώστε να εμφανιστούν περισσότερα ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα στην αγορά. Όταν ας πούμε, μια εταιρεία παρουσιάζει ένα προϊόν το οποίο είναι ενεργειακά αποδοτικότερο από ένα άλλο, φυσικά αυτό αυξάνει τον ε, θεμητό ανταγωνισμό και τις επιλογές των καταναλωτών. Η πολιτική λοιπόν αυτή στέφθηκε με επιτυχία ε, και ε, σε συνδυασμό με τον οικολογικό σχεδιασμό. Εκτιμούμε λοιπόν ότι μέχρι το 2020 η αιτήση εξοικονόμηση ενέργειας ε, ως αποτέλεσμα των πολιτικών αυτών ανέρχεται στην πρωτογενή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της Ιταλίας ανά Και αυτό είναι αναγκαίο έτσι ώστε να φτάσουμε το στόχο του 20% εξοικονόμησης μέχρι το 2020. Αυτή είναι η μία πλευρά του νομίσματος. Η άλλη πλευρά του νομίσματος έχει να κάνει με την τρομερή επιτυχία της πολιτικής αυτής λόγω της υπερπροσφοράς προϊόντων στις ανώτερες κλάσεις. Ε, όταν πηγαίνεις ε, για παράδειγμα να αγοράσει με ένα πλυντήριο θα δεις ότι, ότι πολλά από αυτά είναι α συν, α συν συν και όταν αγοράζεις ε, πολλές φορές με ένα πλυντήριο το οποίο είναι ενεργειακής κατηγορίας α συν υστερεί κατά πολύ σε σχέση με το α συν συν. Γι' αυτό λοιπόν προχωρήσαμε σε μία ανακατάταξη από το 2007 17 Συμφωνήσαμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να γίνουν πιο σαφείς ε, οι κλάσεις αυτές, ε, να μην υπάρχουν λοιπόν αυτά τα συν στο α και η νέα ε, επισήμανση να αρχίζει από το α και να τελειώνει στο g. Η δέσμη μέτρων λοιπόν αυτή αποτελείται από πέντε συστήματα επισήμανσης για τις πιο συχνές ηλεκτρικές συσκευές, ψυγεία, πλυντήρια ρούχων, πλυντήρια πιάτων, φωτισμό και ε, ηλεκτρονικές οθόνες και τηλεοράσεις. Οι εφαρμογές αυτές βρίσκονται, οι συσκευές αυτές έχουν εφαρμογή παντού, μέχρι και σε αυτόματους ε, πολιτές. Επίσης υπάρχουν και άλλα μέτρα οικολογικού σχεδιασμού και εκεί έχουν γίνει αναθεωρήσεις στην ενεργειακή επισήμανση. Έχουμε λοιπόν υποβάλει την ε, έκθεσή μας στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο για εξέταση. Εμείς ε, θα θέλαμε πάρα πολύ να στηρίξετε αυτές τις πράξεις κατά εξουσιοδότηση για τη νέα επισήμανση. Η νέα αυτή επισήμανση θα είναι διαθέσιμη στους ε, καταναλωτές μέχρι την 1η Μαρτίου 2021, εκτός από ε, τον φωτισμό, όπου θα είναι διαθέσιμη ένα χρόνο αργότερα. Αν βλέπετε τις οθόνες θα δείτε τις ε, νέες ε, ετικέτες στα δεξιά σε σχέση με τις παλιές στα αριστερά. Νομίζω πως εδώ υπάρχει περισσότερη σαφήνεια. Δεν θα έχουμε λοιπόν α συν, συν, συν, α συν, συν και α συν. Εδώ θα αδειάσει σταδιακά η κατηγορία Α, λόγω της ανακατάταξης αυτής. Επίσης, είναι πολύ σημαντικό ότι τώρα στην ε, επισήμανση θα υπάρχει ένας κωδικός QR, αυτό που βλέπετε πάνω δεξιά στην ε, δεξιά εικόνα. Ε, σκανάροντας τον κωδικό αυτό θα πηγαίνετε σε μία ειδική σελίδα όπου ο κατασκευαστής θα παρέχει πληροφορίες οι οποίες σταδιακά θα γίνουν προσβάσιμες και για τους καταναλωτές. Θα περιέχονται λοιπόν πληροφορίες για την ε, ηλεκτρική αυτή συσκευή και αυτό θα αυξήσει την ε, διαφάνεια αλλά και ε, την δυνατότητα εφαρμογής της νέας, του νέου συστήματος επισήμανσης για τα κρατημέλη. Θα υπάρχουν 7 νέες κατηγορίες εξοικονόμηση μέχρι 38 τεραβατορών ανά έτος. Το ίδιο δηλαδή με την ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας της Ουγγαρίας. Ελπίζουμε λοιπόν στη στήριξή σας για την ε, πρόταση αυτή, έτσι ώστε να καταφέρουμε να, την, ολοκληρώσουμε τον κύκλο παρουσίασης μέχρι, ε, πάρα πολύ σύντομα. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω τώρα το λόγο στον εισηγητή, εισηγητή κύριο Ταμπουράνο για να μας πει και αυτός δύο λόγια για, το, την πρόταση αυτή. Από το 2015 το επεξεργαζόμαστε. 2019 είμαστε σήμερα, 2021 θα καταφτάσουν αυτές οι ετικέτες. Βήμα πρόδεινα αυτό. Είχαν ξεπεραστεί από τεχνολογία αυτές οι ετικέτες. Αυτή η πρώτη Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσιάζει κάποια όρια. Είναι μια ετικέτα της Ευρωπαϊκής Ενώση που δεν αντιστοιχεί στην τεχνολογία και στο σύγχρονο καιρό. Υπήρχαν δυνατότητες στον κανονισμό που θέλαμε να είναι μελλοντοστραφής ο κανονισμός. Θα μπορούσαμε να προστατεύσουμε τους καταναλωτές έναντι της χρήσεως του, του marketing θα έπρεπε να επεξεταστούν οι παράμετροι και αποδοτικότητα ενεργειακή. Να μην αγοράσουν τεράστιο ε, ψυγείο ε, που είναι κλάση α, ενώ το άλλο ψυγείο είναι σε, μόνο για marketing σε κατηγορία Β. Αυτή, αυτό θέλαμε να το αποφύγουμε, να αγοράζουν οι καταναλωτές μεγαλύτερες συσκευέ από ό,τι χρειαζόταν. Δεν υπάρχει δυνατότητα επίσης ανιχνησιμότητας. Θέλουμε να έχουμε κυκλική οικονομία και χάνουμε μία δυνατότητα που ήδη είχε προβλεφθεί από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Τέλος, πιο σημαντικό, άλλη χαμένη ευκαιρία. Είχαμε ένα clean energy package στην οδηγία για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και για την ηλεκτρική αγορά την οδηγία. Το demand response, ανταπόκριση στη χρήση πλευρά των χρηστών. Θέλαμε να εφαρμοστεί το μέτρο αυτό. Διαχείριση προσφοράς και ζήτησης. Να υπάρχει το Smart Appliance Reading, δηλαδή κάποιες ηλεκτρικές συσκευές θα μπορούσαν να λειτουργούν ή να σβήνουν όταν η ηλεκτρική ενέργεια που αυτοπαράγεται κοστίζει λιγότερο ή περισσότερο. Εύκολη λύση, φτηνή, προσβάσιμη. Αυτές οι έξυπνες συσκευές Smart Appliances δεν παρουσιάστηκε, δεν αναφέρεται. Δεν ξέρω πότε θα φτάσει αυτό. Όλα ανεβλήθησαν για το 2025, 2026. Όταν εκατομμύρια νέοι βγαίνουν στους δρόμους και στρέφονται σε εμά που παίρνουμε τις πολιτικές αποφάσεις για πιο φιλόδοξες πολιτικές και χάνουν την ελπίδα στην πολιτική. Όταν η πολιτική διακυ τη χειρίζεται η αγορά διότι είναι έτοιμοι οι stakeholders να κινηθούν. Η πολιτική δεν δικεί σωστά μέσω στόχων και κανόνων την αγορά για μετάβαση τεχνική, τεχνολογική και κλιματική το το δυνατό, τότε έχουν απόλυτο δίκιο οι νέοι που το βλέπουν. Τους φαινόμαστε σαν ζόμπι εμείς και δεν είμαστε θέση να δώσουμε απαντήσεις. Χρόνια για ένα κομμάτι χαρτί. Σκεφτείτε να πρέπει να ανταποκριθούμε σε πολύ πιο σοβαρέ ε, προκλήσεις που θα αντιμετωπίσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Είμαι βαθύτατα απογοητευμένος από τι κατεξοδότης συμπράξεις. Δεν θα, δεν θα αντιδράσω, δεν θα προβάλλω αντίσταση. Διότι εάν δεν είχαμε λύσει θα είχαμε μεγαλύτερε ζημιέ αν αναβάλαμε την χρήση των νέων ετικετών περαιτέρω. Αλλά αυτό που συμβαίνει με τις ετικέτες δείχνει για μια ακόμη φορά που ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ανίκανη να αντιμετωπίσει τα, προκλήσει τις προκλήσεις του μέλλοντος. Ευχαριστώ. Θέλετε να πείτε λίγα λόγια σαν απάντηση. Καλώς, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κύριε Ταμπουράνο για τα σχόλια σας και ευχαριστώ για το έργο σας επί αυτού του θέματος. Τα εκτιμούμε αυτά που αναφέρατε τώρα. Τα κατανοούμε αυτά που είπατε, τα σημειώνουμε δεόντως. Και εμείς από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα θέλαμε ταχύτερη εφαρμογή, όμως είναι χρονοβόρα αυτά τα πράγματα και η βιομηχανία χρειάζεται κάποιο χρόνο ούτως ώστε να προσαρμοστεί στα νέα συστήματα και οι συσκευές να δοκιμαστούν σύμφωνα με τις νέες κλίμακες και το καθεξής. Θεωρούμε ότι η θέση σε ισχύ και ο χρόνος, η εποχή που θα δείτε αυτές τις ετικέτες στα καταστήματα είναι ο χρόνος ο ταχύτερος, ο πιο σύντομος που μπορούσαμε να καταφέρουμε. Κατανοούμε και αυτό που λέτε για τις ευφυείς συσκευές, είναι κάτι που όλο και περισσότερο θα γίνεται σημαντικό στο μέλλον. Κάναμε διάφορες μελέτες επ' αυτών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά οι μελέτες καταδεικνύουν ότι θα ήταν πρόημο τώρα να συμπεριλάβουμε πληροφορίες για το κατά πόσο κάτι είναι ευφυέ, το βαθμό στον οποίο η συσκευή μπορεί να ανταποκρίνεται στην κατάσταση του δικτύου. Το πλυντήριό σα, να ανάβει όταν υπάρχει πλεόνασμα ηλεκτρική ενέργεια στο δίκτυο. Δεν είμαστε ακόμα σε θέση αυτό να το αναφέρουμε στην ετικέτα με έναν τρόπο που δεν θα είναι αμφισβητήσιμος όσον αφορά τις παρεχόμενες πληροφορίες. Είναι κάτι που θα μας άρεσε. Και μετά ρωτήσατε πότε θα αναμενόταν κάτι τέτοιο. Ο κύκλος κανονικά για την αλλαγή κλίμακα των τικετών είναι περίπου μια δεκαετία. Πρέπει να είναι μακρύ το χρονικό διάστημα. Δεν θέλουμε να προκαλέσουμε σύγχυση στον καταναλωτή με πολύ συχνή αλλαγή της κλίμακας. Αλλά φαντάζεται κανείς, και το θεωρούμε αυτό στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θα μπορούσαμε να έχουμε μια αλλαγή των κανόνων χωρίς να αλλάξουμε την κλίμακα. Συμπεριλάβουμε θέματα που άπτονται της ευφυΐας του συμπίν της συσκευής σε πέντε χρόνια, όχι μετά τη δεκαετία. Βλέπω ότι θέλετε να πατήσετε το κουμπί σας κύριε Πρόεδρε, τελευταίο σημείο. Όσον αφορά τη δυνατότητα επισκευής των συσκευών και την κυκλική οικονομία, αυτό είναι κάτι που η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να αντικατοπτρίζεται καλύτερα στην ετικέτα, γιατί την ώρα δεν είναι εφικτό πιστεύουμε, αλλά αντικατοπτρίζεται στην οικολογικό σχεδιασμό, όπου κάποια θέματα που αφορούν την επισκευασιμότητα, τη διαθεσιμότητα των ανταλλακτικών και τέτοια πράγματα συμπεριλαμβάνονται σαν πληροφορίε στα μέτρα για την οικολογικό σχεδιασμό. Κάνουμε πρόοδο, νέο τομέα και χρειάζεται κάποιο χρόνο για να τα καταφέρουμε, να τα κάνουμε σωστά με έναν τρόπο ο οποίος είναι πραγματικά σε επαφή με τις ικανότητες και τη βούληση της βιομηχανίας. Αυτά και ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε. Πολύ σημαντική καταξιδότηση πράξη. Πάρα πολύ σημαντική. Σας ευχαριστούμε για την ενημέρωση, την παρουσίαση και ευχαριστούμε και τον κύριο Ταμπουράνο, τον εισηγητή μας. Uh, dear friends, let's... Αγαπητοί φίλοι, Πάμε στι ψηφοφορίες, στην ψηφοφορία μάλλον, των κοινών κανόνων για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου. Όπως ξέρετε, στον πρώτο τριμερή διάλογο καταλήξαμε σε προσωρινή συμφωνία με τη Ρουμανική Προεδρία και η Κορεπέρ στις 20 Φεβρουαρίου ε, ενέκρινε την προκαταρκτική συμφωνία στέλνοντας επιβεβαιωτική επιστολή στον πρόεδρο της Ήτρα, τον υποφαινόμενο. Οπότε ας κάνουμε πρώτα μια δοκιμαστική ψηφοφορία για να δούμε αν λειτουργεί το σύστημα. Άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. μάλλον λειτουργεί το σύστημα. Οπότε, ψηφίζουμε για τους κοινούς κανόνες για την εσωτερική αγορά φυσικού αερίου. Ψηφίζουμε με βάση το άρθρο 69F την προσωρινή συμφωνία με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνουμε την προσωρινή συμφωνία. Σας ευχαριστώ θερμά. Και δυστυχώς τελειώσαμε με τις ψηφοφορίες. Μία είχαμε μόνο. Λυπάμαι πολύ. Τι κρίμα. Τι να πω. Λυπάμαι. Μόνο αυτό έχω να πω. Την επόμενη φορά σίγουρα θα είμαι καλύτερος. Σας το υπόσχομαι. Σας υπόσχομαι την επόμενη φορά θα έχουμε τουλάχιστον 20 λεπτά ψηφοφορίες. Σας ευχαριστώ θερμά. Επειδή παρά ήταν σύντομες οι ψηφοφορίες και δεν το ευχαριστηθήκατε, παραμείνετε στην αίθουσα, δεν χρειάζεται να φύγετε για να περάσουμε στο σημείο 5 λέει ο πρόεδρος, όχι το 6-6, που είναι η παρουσίαση από το Γενικό Διευθυντή Μινή Κριστορή, που θα μας παρουσιάσει την οδηγία για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ε, και παρουσίαση σχετικά με την κατεξιοδότηση πράξη. Αλλά πρώτα θα κάνουμε ένα τρίλεπτο διάλειμμα πριν ακούσουμε την παρουσίαση από τον Γενικό Διευθυντή, τον κύριο Ριστορή. Uh, Κύριε Γενική Διευθυντά, εξοδότηση πράξη, πολύ σημαντική για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Σχετική οδηγία. Θα ήθελα να πω ότι η οδηγία για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ε, εγκρίθηκε το Δεκέμβριο του 2018 και εξουσιοδοτεί την Επιτροπή να υιοθετήσει την κατεξοδότηση πράξη μέχρι την 1η Φεβρουαρίου του 2019 θεσπίζοντας κριτήρια για την πιστοποίηση ε, μικρής έμεσης ε, χρήσης γης ε, και αλλαγής χρήσης γης, ε, ε για τα βιοκαύσιμα, βιο... καύσιμα, βιομάζα, καύσιμα από βιομάζα και για να ε, προσδιοριστεί ο μεγάλος κίνδυνος άμεσης ε, χρήσης γης και αλλαγής χρήσης γης ε, με διεύρυνση της έκτασης παραγωγής σε γη με υψηλή δεσμευσή και αποθεμάθρακα. Στις 8 Φεβρουαρίου η Επιτροπή εξέδωσε το σχέδιο κατεξοδότηση πράξης, ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις που κράτησαν ένα μήνα και τώρα ήρθε η σειρά σα να μα παρουσιάσετε αυτή την κατεξοδότηση πράξη στην Επιτροπή μα, κύριε Γενική Διευθυντά. Κύριε Πρόεδρε, αξιότιμοι Ευρωβουλευτέ, θα ήθελα καταρχήν να εκφράσω την αγνωμοσύνη μου για τις πολύ επικοδομητικές ε, συζητήσεις που είχαμε με πολλούς ευρωβουλευτές κατά την εκπόνηση αυτής της κατεξοδότησης πράξης. Θα σας παρουσιάσω την προσέγγιση μας κατά την υθέτηση αυτής της κατεξοδότηση πράξης και θα σας πω πόσο επηρεαστήκαμε και λάβαμε υπόψη ε, τα σχόλια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και τις δημόσιες Διαβουλεύσης που είχαμε. Καταρχήν να θυμηθούμε το πλαίσιο. Έχουμε την αναθεώρηση οδηγία για την προώθηση της χρήσης ενέργειας από νεώσιμε πηγέ ε, που ενέκνε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Συνομοθέτης να ευχαριστήσω εδώ και το Κοινοβούλιο, τον Ζουζέ Μπλακον Λόπες, τον εισηγητή, αλλά και τον κύριο Εκχόουτ από την Επιτροπή Περιβάλλοντος. Η αναθεωρημένη λοιπόν οδηγία ήδη προβλέπει όλα τα απαραίτητα κριτήρια για την προσέγγιση της, ε, του υψηλού κινδύνου για τα βιοκαύσιμα προκειμένου να τηρηθούν οι στόχοι μας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Η οδηγία απαιτεί τα εξής. Για με ψηλής ενέργειας προβλέπεται το πάγωμα για την περίοδο 2021-2023 σε εθνικό επίπεδο από το, το 2019 και θα έχουμε μια σταδιακή εγκατάλειψη, μείωση που ξεκινάει από τον Ιανουάριο του 2024 και θα ολοκληρωθεί το αργότερο αυτή η κατάργηση το 2030 με μια σταδιακή μείωση. Επίσης υπάρχει εξαίρεση για χαμηλού ελέγχου, ε, ε, χαμηλού κινδύνου βιοκαύσιμα. Και ζητήσατε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να θεσπίσει τα κριτήρια για την προσέγγιση αυτή και να σας ενημερώσει ε, για το αποτέλεσμα των προσπαθειών τη. Ποια είναι τώρα η προσέγγιση που υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην κατεξοδότηση πράξη. Και για τον υψηλό και τον χαμηλό κίνδυνο. Καταρχήν τα βιοκάψιμα τα ξυνομούνται ως ψηλού κίνδυνο α με βάση τα εξής σωρευτικά κριτήρια. Ε, αύξηση της ελάχιστης επέκτασης της, αγοράς, της ε, έκτασης παραγωγής με πάνω από 10% ε, επέκταση με, σε μια περιοχή που θα έχει μεγάλο απόθεμα άνθρακα. Τώρα, τι συνιστά σημαντική επέκταση. Το 10% είναι το ποσοστό που επιλέξαμε, προκειμένου όλα τα βιοκαύσιμα που συμπεριλαμβάνονται στο στόχο για τις ΑΠΕ να μας οδηγούν σε σημαντική εξοικονόμηση καυσέριων και να περιορίσουμε την απώλεια σε γεές με υψηλή βιοπικιλότητα. Είναι επίσης σημαντικό να, ε, να πούμε ότι το φινικέλο εμπίπτει σε αυτό το high risk feedstock. Δεύτερο σωρευτικό κριτήριο για την πιστοποίηση ε, βιοκαυσίμων χαμηλού κινδύνου. Καταρχήν θα πρέπει να υπάρχει συμμόρφωση με το κριτήριο βιωσιμότητας, χρήση των επιπλέον ε, ζωοτροφών ε, από την ήδη χρησιμοποιημένη, ε, χρησιμοποιημένη γη και λήψη υπόψη του στόχου της βιοποικιλότητας. Και τέλος, η κατεξόδηση πράξη Ευρωπαϊκής Επιτροπής λαμβάνει υπόψη κυρίως τις σημαντικές παρατηρήσεις και τα σχόλια που μα έστειλε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αλλά και άλλοι συμφεροντούχοι και εκπρόσωποι της κοινωνία των πολιτών από τι δημόσιε διαβουλεύσει. Σε τρία επίπεδα έλευσαν υπόψη οι παρατηρήσει σε ό,τι αφορά την εξαίρεση για τους μικροκαλλιεργητές. Ε, θωρακίζουμε τον ορισμό ώστε να μην επιτρέπονται απάτες. Είναι θωρακισμένος από απάτες και έχουμε το, κατόφλι που περιορίζεται στα 2 εκτάρια. Η επιλογή των 2 εκταρίων ε, είναι το σχόλιο που μας έδωσαν ε, οργανώσεις τροφίμων και γεωργίας. Επίσης, οι μικροκαλλιεργητές θα πρέπει να πληρούν το κριτήριο της βιωσιμότητας και θα πρέπει να αυξήσουν την παραγωγικότητά τους για να είναι επιλέξιμοι. Δεύτερον, εξαίρεση για τις ζωοτροφές που ε, για τις πρώτες ύλες που προέρχονται από μη χρησιμοποιημένη γη. Κάτι τέτοιο ε, δικαιολογεί εξαίρεση σε περίπτωση που έχουμε υπερβεί το οικονομικό κριτήριο. Και τρίτον, πιστοποίηση, διαδικασία πιστοποίησης που ενισχύθηκε ε, χάρη στην ενίσχυση του ελέγχου και του κριτηρίου της διαφάνειας. Επίσης, ε, διευκρινίστηκε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα θεσπίσει αναλυτική διαδικασία στην κατεξουδότηση πράξη, όπως απαιτείται στο άρθρο 30 της οδηγίας, πριν τα τέλη Ιουνίου του 2021. Εγκατακλείδη. Ε, καταλήξαμε σε μια ισορροπημένη εύρωστη προσέγγιση που στηρίζεται σε αξιόπιστα δεδομένα και πορίσματα. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συνεχίσει να παρακολουθεί όλες τις εξελίξεις και το αργότερο μέχρι τις 30 Ιουλίου 2021 θα αξιολογήσει και τα τελευταία επιστημονικά κριτήρια και εν ανάγκη θα προτείνει τροποποίηση της προσέγγισης. Άλλωστε, για το 2023 προβλέπεται ήδη αξιολόγηση και αναθεώρηση ενδεχομένω οδηγία. Και είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη όλοι αυτοί οι παράμετροι και η σωστή διαχείρισή του. Γιατί το θέμα είναι ευαίσθητο, όπω ξέρετε. Και έχουμε και την αντίδραση πολλέ φορέ χώρε παραγωγή. Αλλά κάναμε την επιλογή της βιωσιμότητας και είναι σημαντικό να εμείνουμε σε αυτήν και να την εφαρμόσουμε σωστά και να πείσουμε ε, τους εταίρους μας και παγκοσμίω ώστε να στραφούν ε, σταδιακά προς τη δική μας κατεύθυνση που είναι η βιωσιμότητα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ο κύριος Μπλάνκο Λόπες, ο εισηγητής, έχει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα Πρώτα απ' όλα να επισημάνω την ανάγκη της κατεξουδότης πράξη που συμπληρώνει την οδηγία για τις ΑΠΕ προκειμένου να έχουμε τα κριτήρια που διέπουν τα βιοκαύσιμα υψηλού χαμηλού κινδύνου σε ό,τι αφορά την αλλαγή της γης. Ε, ήταν πολύ σκληρές οι διαπραγματεύσεις ε, για το θέμα αυτό και χρειάστηκε να τις διεκπαιρεώσουμε για να σώσουμε την οδηγία. Τελικά καταλήξαμε σε μια ορθολογική συμφωνία, ισορροπημένη και περιμέναμε και την κατεξοδότηση πράξη για τη συμπλήρωση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζουμε ότι είχε ελάχιστο χρόνο για να ανταπεξέλθει σε αυτή τη σημαντική πρόκληση και να βρει λύσει για να λάβει μια απόφαση ε, ό,τι αφορά την αλλαγή τη χρήση γη για την παραγωγή βιοκαυσίμων πρώτη γενιά και ήδη βιοκαυσίμων που επηρεάζουν την αποψήλωση, τις ε, εκπομπές, την απασχόληση και έχουμε και το θέμα της ανταγωνιστικότητάς μας διεθνώς. Ε, στο προσχέδιο είχαμε αρκετές αδυναμίες, παραθυράκια και κερκόπορτες που υπέσκαπταν όλο το έργο που είχαμε κάνει και υπονόμευαν το έργο μας για να ε, αξιοποιήσουμε τη βιοενέργεια βιώσιμα. Πάντως αναγνωρίζουμε το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή την και σε εμά, στην Επιτροπή μας και στους συμφεροντούχους, γράστηκε τα αιτήματά τους, περιόρισε τα κενά, διευκρίνησε τα κριτήρια και τους ορισμούς και εξήγησε καλύτερα το πεδίο εφαρμογή της κατεξοδότησης πράξης. Βέβαια, όπως λέμε, το τέλειο είναι εχθρός του καλού. Ως εκ τούτου, παρά τις κριτικές που ασκούμε στην κατεξοδότηση πράξη, παρόλο που ε, υπάρχουν ακόμα κάποιες αδυναμίες, θα πρέπει να το δούμε με τη σωστή απόσταση και να αναγνωρίσουμε την σωστή κατεύθυνση για τις ΑΠΕ. Ε, άλλωστε, αν απορρίψουμε αυτή την κατεξοδότηση πράξη, θα βρεθούμε σε πολύ χειρότερη θέση και θα έχουμε ένα μεγάλο χρονικό ορίζοντα χωρίς κριτέρια ε, για τα βιοκαύσιμα με μεγάλο κίνδυνο για αλλαγή χρήση γη. Και δεν θα μπορέσουμε να έχουμε θετικά αποτελέσματα. Πιστεύω ότι με αυτή την κατεξοδότηση πράξη σημειώνουμε πρόοδο για τη βιώσιμη χρήση της βιοενέργειας και κάνουμε ένα πολύ σημαντικό βήμα για να μειώσουμε την αποψήλωση των δασών, να μειώσουμε και τα καυσαέρια. Η βιώσιμη πραγματικά βιοενέργεια είναι απολύτως απαραίτητη για να επιτύχουμε την ουδετερότητα σε ό,τι αφορά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Γι' αυτό θα ήθελα να, συστήσω, να σας συστήσω την έγκριση αυτής της κατεξοδότησης πράξης. Σας ευχαριστώ πολύ για τα σχόλια. Θα δώσω τώρα το λόγο στον κύριο Λάγκεν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γενική Διευθυντά. Σας καλωσορίζουμε για την... Ε, που στην Επιτροπή και σας ευχαριστούμε για την παρουσίαση. Φυσικά η βιωσιμότητα έχει κινδύνους και η πιστοποίηση είναι και μία λύση. Βέβαια, αυτό που δεν καταλαβαίνω είναι αυτή η μονομερής απαγόρευση του φινικέλαιου. Το φινικέλαιο είναι 10 φορές πιο αποτελεσματικό στην κατασκευή βιοκαυσίμων από... σε σχέση με τα υπόλοιπα. βιοκαύσιμα που παράγονται από άλλα έλαια. Η Ινδονησία και η Μαλαισία είναι οι χώρες που έχουν το 95% της παγκόσμιας παραγωγής φινικέλαιου. Στην Ινδονησία η παραγωγή μοιράζεται σε 400.000 παραγωγούς. Στη Μαλαισία είναι ακόμα ε, περισσότεροι. Αυτό ε, δείχνει πόσο σημαντικό είναι το φινικέλαιο. Βλέπουμε τώρα πως ε, θέλει να εισαχθεί αυθαίρετα ένα ανώτατο όριο, όμως χρειάζεται να δώσουμε την ευκαιρία και στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Πιστοποίησης να δείξει την αξία του. Τώρα, στη Μαλαισία. Σίγουρα αποψηλώνονται μεγάλε εκτάσει για την ε, καλλιέργεια φινικελαίου. Όμως οι παραγωγοί ανήκουν σε διάφορες ε, ενώσει και ο κάθε παραγωγός έχει μικρή έκταση γη στην οποία καλλιεργεί. Ε, το θέμα της βιωσιμότητα λοιπόν πρέπει να το δούμε σφαιρικά, να το δούμε και από τις δύο πλευρές. Φυσικά και στηρίζω την βιωσιμότητα, Όμω από την άλλη το γεγονός ότι η γαλλική κυβέρνηση αποφάσισε να απαγορεύσει το φινικέλαιο δεν θα πρέπει να επηρεάζει την ευρωπαϊκή πολιτική. Βλέπουμε ότι προσπαθεί να γίνει το ίδιο και με τη σόγια. συζητάμε για το πόσο ακατάλληλη είναι η σόγια σε κάποιες περιπτώσει και τώρα βλέπουμε ότι θέλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να χορηγήσει μια εξαίρεση για τη χρήση σόγια σε ζωοτροφές. Μετά, από την άλλη, δείτε τι γίνεται και στην άλλη πλευρά του Ολλανδικού, στην ε, Βραζιλία, που αποψηλώνονται τεράστιες ε, δασικέ ε, εκτάσει. Και τώρα ασχολούμαστε με δύο αναπτυσσόμενες ε, χώρες και το Φινικέλαιο. Και μην ξεχνάτε πως αυτές οι δύο χώρες ε, κατέχουν το 95% της παγκόσμιας παραγωγής ε, Φινικέλαιο. Νομίζω πως αυτή η πρόταση δεν είναι λοιπόν κατάλληλη. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο, Ο κύριος Μαρτάν, Εντουάρτ Μαρτάν έχει το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Δεν θα μακρηγορήσω. Ακόμα και αν το κείμενο έχει βελτιωθεί σε σχέση με το αρχικό, αλλά καταρχήν κατά της εκμεταλλεύσεως του φινικελαίου. Το είπα και την περασμένη φορά. Ας έχουμε εμπιστοσύνη στη βιομηχανία. Ακόμα και αν έχει βελτιωθεί αυτό το κείμενο, θα μπορέσουν αυτοί να οργανωθούν και θα ξεπεράσουν τα εμπόδια που θα τους βάλουμε. για να μην εξελιχθούν τα πράγματα όσον αφορά την μαζική εκμετάλλευση του φινικελαίου που θα δημιουργούσε προβλήματα τα δάση. Ε, γίνανε γιγαντιές διαδηλώσεις των νέων στον κόσμο και μας κατηγορούν ότι δεν προσέχουμε την αλλαγή του κλίματος και τη θέρμανση του πλανήτη. Αυτή η νέα γενιά λέει με έναν τρόπο αρκετά ομό ότι πρέπει να σακου... και θέλουν να ακουστούν ότι εμείς οι παλιοί δεν νοιαζόμαστε για το πλανήτη γιατί θα πεθάνουμε σύντομα όλοι. Αυτά άκουσα χτέ σε αυτά που λέγανε οι νέοι. Μήπως δεν έχουμε εμείς υποχρέωση να διαφερθούμε και εμείς για το θέμα αυτό του πλανήτη, για οποιοδήποτε λόγο. Να μου απαντήσετε σε μια ερώτηση. Γιατί έχουμε αυτή την εξαίρεση, εξηγήστε μας. Ποια είναι η βάση της εξαίρεσης για να δεχθούμε το φινικέλαιο, έστω και από μικρές εκμεταλλεύσεις αν παράγεται. Και δεν θα να μιλήσω. Θα με αφήσει να μιλήσω ή όχι. Θα γίνει. Να γελάτε στο τσίρκο σας εσείς. Άντε. Άντε μπράβο. Εγώ θα ήθελα να μου απαντήσετε σε αυτή την ερώτηση. Γιατί αυτή η θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Τι είναι. Περί πρόκειται. Τι είναι. Πιέσεις από πλευράς Μαλαισίας κλπ. Για πωλήσει όπλων, για να αγνοηθούν πωλήσει όπλων όπως ε, Ραφάλ κλπ. Ευχαριστώ. Είμαστε ανοιχτοί, λέει ο Πρόεδρος, για κάθε ερώτηση. Αν κάποιος επιθυμεί να ξαναπάρει το λόγο, και αυτό είναι δυνατόν. Δεν έχω μακροσκελή κατάλογο μιλήτων, βλέπετε. Η κυρία Γκρίφιν, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ. Γέρτζη, χαίρομαι που σε βλέπω εδώ, Ντομινίκ. Θέλω να στηρίξω αυτά που είπε ο Ντουάρτ. Η δουλειά που κάναμε όσον αφορά το πακέτο για την καθαρή ενέργεια για όλους τους Ευρωπαίους πολίτες, βάζοντας τους πολίτες στο επίκεντρο της Ενεργειακής Ένωσης δεν ξέρω, δεν βλέπω να έχει νόημα αυτή η εξαίρεση για το φινικέλαιο. Η ερώτησή μου είναι ίδια όπω αυτή του Εντουάρ. Γιατί ξυλώνουμε την καλή δουλειά που κάναμε. Την κάναμε συλλογικά. Ε, όλοι συμμετείχαν, όλες οι αντιπροσωπείες, όλες οι πολιτικές ομάδες συμμετείχαν, συνεργαστήκαμε. Προσπαθήσαμε να εξασφαλίσουμε ότι θα σώσουμε τον πλανήτη για τους νέους μας. Να σου πω Γεζή, στο Λίβερπουλ την Παρασκευή υπήρχαν εκατοντάδες, εκατοντάδες, εκατοντάδες νέοι που βγήκαν στους δρόμους και διαδήλωναν για το μέλλον του πλανήτη τους. Θέλω να υποστηρίξω από βρετανικής πλευράς, από βρετανικής αντιπροσωπείας όλα όσα είπε μόλις τώρα ο Εντουάρ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κ. Λάγκεν. Ήθελα να πω πως, ε, εντάξει δεν ήθελα να διακόψω τον ε, αλλά ρωτήσατε πού βρίσκονται αυτές οι εξαιρέσεις για τα δύο εκτάρια, για τους μικρούς παραγωγούς στην Ινδονησία και την ε, Μαλαισία, πώς δικαιολογούνται αυτές οι εξαιρέσεις. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω πώς, ε, στο, πού βασίζεται η γενικότερη εξαίρεση για τη σόγια. Βλέπουμε ότι 21 εκατομμύρια εκτάρια είναι εκτάσεις όπου καλλιεργείται σόγια. Εκεί δεν θα έπρεπε να υπάρξει μια αλλαγή, μια μείωση. Βλέπουμε ότι αυξάνονται συνεχώς οι εκτάσεις όπου καλλιεργείται σόγια. Ε, αλλά χρειάζεται, θεωρώ, πιστοποίηση μεν, ε, κριτήρια βιωσιμότητας, ε, όχι όμως απαγόρευση. Νομίζω πως ε, αν εφαρμοστούν αυστηρά κριτήρια επιλεξιμότητας, βιωσιμότητας, τότε θα έχουμε θετικά αποτελέσματα. Αλλά δεν πρέπει να στερήσουμε από τους αγρότες αυτά τα, αυτή την σημαντική πηγή εσόδων. Μάλιστα. Άλλος κανείς θέλει το λόγο παρακαλώ. Ουδής. Οπότε κύριε Γενική Διευθύντα έχετε το λόγο εσείς. Βλέπετε, τη συζήτηση ήταν πολύ ζωηρή, γιατί το θέμα είναι φλέγον. Ξέρετε, δεν είναι καθόλου εύκολο το ζήτημα αυτό. Θα ήθελα να πω ότι είναι αδύνατο να εντοπίσουμε σε διεθνές επίπεδο άλλη ε, μεγάλη οικονομική ζώνη που να αναπτύσσεται τόσο σημαντικά ε, και να αναπτύσσει τέτοιο κανονιστικό και ρυθμιστικό πλαίσιο υπέρ ε, του πακέτου καθαρής ενέργειας. Όλους τους ανταγωνιστές μας και αν εξετάσετε, βλέπετε ότι εμείς είμαστε μοναδικοί και πρωτοστατούμε. Είμαστε η πιο προηγμένη περιοχή σε ό,τι αφορά το αποτύπωμά μας ενός στιβαρού ρυθμιστικού και κανονιστικού πλαισίου υπέρ τη καθαρή ενέργεια. Και γι' αυτό ακριβώ με τη δική σα υποστήριξη, με την αρρωγή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, καταλήξαμε σε νέου φιλόδοξου στόχου και συμφωνήσαμε σε φιλόδοξε διατάξει και για την οδηγία για τη ΑΠΕ και για την οδηγία για την ενεργειακή απόδοση και για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων και για την οδηγία για την ε, διακυβέρνηση την ενεργειακή διακυβέρνηση, αλλά και όλε τι πτυχέ του οικολογικού σχεδιασμού. Νομίζω ότι όλα αυτά συνιστούν ένα πολύ στιβαρό κανονιστικό πλαίσιο. Δεύτερον, το όραμά μα, όπω ξέρετε, συνδυάζει την ανταγωνιστικότητα με την βιωσιμότητα, την αηφορία. Θεωρούμε ότι είναι εφικτό ο συνδυασμό των δύο στόχων. Και στο πρόσφατο παρελθόν, από το 1990 μέχρι το 2017, το ΑΕΠ μας στην Ευρώπη αυξήθηκε κατά 56% και, ταυτόχρονα μειώσαμε κατά 22% τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου και είμαστε οι μόνοι με τέτοιες υψηλές επιδόσεις παγκοσμίω. Τώρα, για να απαντήσω στα επιμέρους σχόλια. Καταρχήν ευχαριστώ τον εισηγητή, τον κύριο Μπλάνκο Λόπες. Όντως, λάβαμε υπόψη πολλά σχόλια το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Προκειμένου να βελτιώσουμε το σχέδιο της της πράξη. Και κυρίως ό,τι αφορά τα τρία σημεία που σα ανέφερα, Του μικροκαλλιεργητέ, τη μη χρησιμοποιημένη γη και την πιστοποίηση. Σε αυτού του τρει τομεί λάβαμε υπόψη τα σχόλια του Κοινοβουλίου και προσπαθήσαμε να θωρακίσουμε το σύστημα ώστε να αποτρέψουμε τις απάτες, να τις αποφύγουμε και να μείνουμε ε, επικεντρωμένοι στην βιωσιμότητα. Και φυσικά ο στόχος είναι ο περιορισμός της αποψήλωσης των δασών. Και μπορώ τώρα να μεταβώ στο σχόλιο του κυρίου Λάγκεν. Γιατί είχαμε επαφή και με χώρες παραγωγούς, μόνιμη επαφή. Επισκεφθήκαμε την Ιδονησία, τη Μαλαισία και διαπίστωσα με ιδιαίτερη χαρά ότι παρά κάποιες συμπεμονωμένες αντιδράσεις, η Μαλαισία για παράδειγμα συμφώνησε και αποφάσισε να συμπεριλάβει και αυτή τη βιωσιμότητα. Η Μαλαισία αποφάσισε να προστατεύσει τα δάση από την αποψήλωση όσο μπορεί. Και θα πρέπει να εξηγήσουμε σωστά το κείμενό μας. Γιατί όπως ξέρετε και αυτό ισχύει και για τον κύριο Μαχτά και για την κυρία Γκρίφιν, αντιμετωπίζουμε παγκόσμιες προκλήσεις. Είναι σημαντικό λοιπόν να πρωτοστατήσουμε στον αγώνα κατά των κλιματικών αλλαγών. Ταυτόχρονα όμως γνωρίζουμε ότι για να λύσουμε ε, τις προκλήσεις, για να ανταπεξέλθουμε στις προκλήσεις, θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και τους άλλους ανταγωνιστές μας, να προσετερήσουν τη θέση μας. Είμαστε πάνω από το 90% της παρέμβασης. Θα πρέπει λοιπόν να πείσουμε τους διεθνείς μας εταίρους να ε, ασπαστούν και αυτή την βιωσιμότητα και ελπίζω να τα καταφέρουμε, να τους μεταπίσουμε. Νομίζω ότι με την αλλαγή της ε, κατεξοδότηση πράξη έχουμε πολύ συνεπή και συνεκτικά κριτήρια. Και με βάση αυτά τα κριτήρια το φινικέλαιο θεωρείται υψηλού κινδύνου για αλλαγή χρήση γης. Οπότε, δεν θα λάβουμε υπόψη το θέμα αυτό στο πλαίσιο των στόχων ΑΠΕ. Ταυτόχρονα θα πρέπει να συνεχίσουμε το διάλογο με τις χώρες αυτές για να εξηγήσουμε το επιχείρημά μας. Τίποτα δεν είναι μοιραίο. Δεν είμαστε μοιρολάτρες. Θα πρέπει να βρούμε τη σωστή διαχείριση για να ανοίξουμε νέους διόδους στην βιωσιμότητα. Αυτό είναι πολύ σημαντικό για μας. Και επίσης θα ήθελα να σας πω ότι αν είχαμε μια διαφορά μεταξύ φινικελαίου και σόγιας, η διαφορά οφείλεται στις αντικειμενικές ε, διαπιστώσεις που κάναμε με βάση την επίπτωση που έχουν αυτά τα δύο προϊόντα στις διάφορες επιφάνειες ε, και στα δάση. Και η ανάλυση κατέληξε τεράστιες διαφορές μεταξύ του φινικελαίου και της σόγιας ως προς επιπτώσεις. Και γι' αυτό προς το παρόν το φινικέλο το κατατάξαμε στα βιοκαύσιμα υψηλού κινδύνου για την αλλαγή χρήσης γης. Γιατί 47% δίνει ε, το ποσοστό για το φινικέλο, είναι 8% μόνο για τη σόγια. Και όλα αυτά στηρίζονται σε αντικειμενικά στοιχεία και σε αξιόπιστα στοιχεία. Δεν θέλουμε να εθελοτυφλούμε στην κατάσταση άλλων χωρών. Απλώς θέλουμε να έχουμε θετικό διάλογο μαζί τους και σε αυτό να δώσουμε έμφαση. Είχαμε συνεχή διάλογο και με τις χώρες αυτές για να εξηγήσουμε τους λόγους των επιλογών μας. Κάναμε τις επιλογές αυτές όχι για να προκαλέσουμε ένα Big Bang, μια κοσμογονική έκρηξη, αλλά ε, μια σταδιακή μείωση μέχρι την κατάργηση και λαμβάνοντας υπόψη τα ισχύοντα στοιχεία. Αυτό ζητάει η οδηγία. Με μια περίοδο παγώματος μεταξύ του 2021 και του 2023 και μια σταδιακή μείωση, ένα phasing out που λέμε, μεταξύ του 2024 και 2030 το αργότερο. Αυτή είναι λοιπόν, αυτό ήταν ο μύθο τη Αριάδνη που ακολουθήσαμε, αυτή ήταν η κατευθυντήρια γραμμή και κάναμε ό,τι μπορούσαμε ώστε στις εξαιρέσει να συμπεριλάβουμε και κάποιες παραμέτρους για να αποφύγουμε τις καταχρήσεις και τις απάτες και να αποφύγουμε ακριβώς αυτό που είπατε, ε, την παράκαμψη της νομοθεσίας. Θέλουμε να αποφύγουμε παράκαμψη της νομοθεσίας και γι' αυτό θα έχουμε ένα σύστημα πιστοποιημένο και αναγνωρισμένο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μας δίνει πολύ ξεκάθαρα στοιχεία ελέγχου. Ο, έλεγχος, ο αξιόπιστος έλεγχος πιστοποίησης θα οδηγήσει και στην αξιοπιστία του συστήματος. Και γι' αυτό βάζουμε τα δυνατά μας για να εξασφαλίσουμε μια αποτελεσματική και συνεπή διαχείριση του συστήματος. Ευχαριστώ. Thank Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Γενική Διευθυντή. Ήταν πολύ επικοδομητική η ανταλλαγή απόψεων. Και είναι υποχρέωσή μας εξάλλου να συζητάμε τόσο σημαντικά θέματα που αφορούν και τις ε, εξουσιοδότηση πράξης. Θα περάσουμε τώρα στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης. Ενημέρωση Λοιπόν, για τις αποστολές της Ήτρε. η πρώτη ενημέρωση έχει να κάνει με την 13η Σύνοδο του Φόρουμ για τη Διακυβέρνηση του Διαδικτύου στο Παρίσι από τις 12 ως τις 14 Νοεμβρίου 2018. Ήταν παρόντες ορισμένοι συνάδελφοι, μέλη της ε, Επιτροπής, όπου συζητήθηκαν θέματα κυβερνασφάλειας, ε, τεχνολογίας και του Κέντρου Δεξιοτήτων. Ξεκίνησαν διαπραγματεύσεις πριν από λίγες μέρες και τα αποτελέσματα ήταν ε, απροσδόκητα καλά. Η συγγήτρια Χιούλια Ρέντα είναι εδώ η οποία θα μας ενημερώσει. Ε, δεν βλέπω κάποιον άλλο συνάδελφο να είναι ε, παρόν. Νομίζω λοιπόν πως θα μας ενημερώσετε για όσα συζητήθηκαν. Έχετε λοιπόν το λόγο. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ναι, συμμετείχα στην αποστολή στο Παρίσι, στο Φόρουμ Διακυβέρνηση του Διαδικτύου. Με χαρά μου λοιπόν θα σα ενημερώσω, αλλά και θα σα ενημερώσω και για το, τα αποτελέσματα του τριμερού διαλόγου για το Κέντρο Κυβερνασφάλεια. Ε, Απέστα λοιπόν η αποστολή μα ε, στο Φόρουμ Δικυβέρνηση του Διαδικτύου. Η επιτροπή μα ήταν η καθήλυνα αρμόδια μαζί με τι επιτροπέ πολιτισμού, ΙΝΚΟ, Γιουρί και ΛΥΜΠΕ, αλλά και το, ε, πάνελ. Συμμετείχαμε λοιπόν στον, ε, στο φόρουμ για τον διάλογο σχετικά με τη διακυβέρνηση του διαδικτύου. Πάνω από 200 συμμετέχοντες παρευρέθησαν στο Παρίσι. Είχαμε λοιπόν πολύ μεγάλη συμμετοχή. 171 συνεδρίες έλαβαν χώρα για θέματα όπως η κυβερνασφάλεια, η εμπιστοσύνη, η ιδιωτικότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και άλλα εκτός από τη συμμετοχή μας στο επίσημο πρόγραμμα ως αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είχαμε και αρκετές διμερείς συναντήσεις. Η αντιπροσωπεία λοιπόν του Κοινοβουλίου συναντήθηκε με το Φόρουμ Διακυβέρνηση Νεολαία για να συζητήσει θέματα όπω ο φοβισμό στο διαδίκτυο, οι ψευδεί ειδήσει, αλλά συναντηθήκαμε και με εκπροσώπους κοινωνία των πολιτών για να συζητήσουμε ε, τις ε, πιθανέ μελλοντικέ μεταρρυθμίσεις Συναντηθήκαμε και με τη Eurodic για να συζητήσουμε την συνεργασία μεταξύ Ευρωβουλευτών και του Διεθνούς Φόρουμ, αλλά και τον ε, ρόλο μας ε, στις ε, μελλοντικές εξελίξεις. Επίσης, συναντηθήκαμε με τον αναπληρωτή Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Εμπορίου των Ηνωμένων Πολιτειών για να συζητήσουμε θέματα κυβερνασφάλειας, ουδετερότητας του διαδικτύου και συλλογής δεδομένων. Συζητήθηκαν επίσης θέματα του απορρίτου των ε, δεδομένων, πλαστογράφησης, αλλά και την ανάγκη καλύτερης εκπαίδευσης και κατάρτισης των ε, τελικών χρηστών του διαδικτύου. Επίσης, συζητήσαμε και συναντηθήκαμε με διάφορους ε, φορείς σχετικά με την ελευθερία της έκφρασης στο διαδίκτυο, την παρεμβολή στη διαδικασία εκλογών, και ανταλλάξαμε απόψεις με πάρα πολλούς ε, λοιπόν ε, φορείς, ε, διότι το φόρουμ ακριβώς αυτόν τον ρόλο έχει να φέρνει κοντά εκπροσώπους από κάθε γωνιά του κόσμου και από κάθε χώρα του πλανήτη. Η επόμενη συνάντηση θα γίνει στο Βερολίνο από τις 25 έως τις 29 Νοεμβρίου 2019. Και κύριε Πρόεδρε, αν θέλετε μπορώ να προχωρήσω αμέσως στην ενημέρωση για το επόμενο σημείο, εκτός αν υπάρχει κάποιο σχόλιο για το Φόρουμ Διακυβέρνηση του Διαδικτύου. Ναι, υπάρχει κάποιο σχόλιο λοιπόν, κάποια ερώτηση για την αποστολή μας στο Παρίσι. Σχετικά με το Φόρουμ Διακυβέρνησης του Διαδικτύου. Δεν βλέπω κάποιο σχόλιο, οπότε λοιπόν μπορείτε να προχωρήσετε στο επόμενο θέμα για το οποίο είστε εισηγήτρια. Ναι, θα σας ενημερώσω λοιπόν για τα αποτελέσματα του πρώτου τριμερούς διαλόγου για το κέντρο δικτύωσης και ε, δεξιοτήτων στον κυβερνοχώρο. Ήταν ο πιο γρήγορο τριμερής διάλογος ε, στην ιστορία. Έγινε επίσης την ε, Τρίτη όπου εγκρίθηκαν θέσει τόσο του Κοινοβουλίου όσο και του Συμβουλίου. Στόχο μα ήταν να επιτύχουμε μια μερική διαπραγματευτική εντολή πριν τη λήξη τη κοινοβουλευτική θητεία. Το θέμα αυτό περιλαμβάνει και στοιχεία για αφορούν το πολιτέ δημοσιονομικό πλαίσιο, τα οποία έχουν πει σε ε, επανενθέσεις αυτά θα αλλάξουν, όμως προσπαθήσαμε να ολοκληρώσουμε τις διαπραγματεύσεις εντός της ε, θητείας μας για όσο το δυνατόν περισσότερα θέματα. Το ζητούμενο είναι το ποιον ρόλο θα έχει η Ευρωπαϊκή Ένωση στο κέντρο κυβερνασφάλειας, ε, τι θα πρέπει να επενδύσει και ποια θα είναι ε, τα καθήκοντά του. Συζητήθηκαν και οι εγκαταστάσεις ε, του και θεωρώ πως είναι σημαντικό το κέντρο αυτό να εφαρμόζει μια κοινή ευρωπαϊκή στρατηγική για την ασφάλεια στον χώρο και όχι απλά να χρηματοδοτεί εθνικά project. Είναι μια θέση την οποία θα υπερασπιστούμε στον ερχόμενο τριμερή διάλογο. Όμως αυτό που χρειάζεται είναι αρκετή ευελιξία από πλευρά Συμβουλίου έτσι ώστε να σημειώσουμε πρόοδο πριν την λήξη τη κοινοβουλευτική μα θητεία. Ευχαριστώ. Την επόμενη εβδομάδα ή αργότερα θα ολοκληρωθεί ο τριμερής διάλογος στο Στρασβούργο ενδεχομένως. Ίσως θα καταφέρουμε. Ερώτηση ουδεμία. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία μου. Ευχαριστώ Γιούλια. Επόμενο σημείο. Σημείο 8. Αποστολή της Ήτρες στο Ισραήλ. Ο κύριος Πολ Ρούμπικ, επικεφαλής αντιπροσωπείας, θα είναι εδώ σε μισή ώρα. Θα το συζητήσουμε λοιπόν αργότερα. Τώρα, πάμε στο σημείο 9. Αποστολή της Ήτρες στη Σουηδία. 27 Φεβρουαρίου με 1η Μαρτίου φέτος. Ο κ. Φέντερλε ήταν επικεφαλής της αντιπροσωπείας. Ο συνάδελφος Γιάκοπ Νταλουγκέ από τους Πρασίνους είναι εδώ, που ήταν και αυτός στην αποστολή. Θα μπορούσατε να μας δώσετε κάποιες πληροφορίες για την αποστολή στη Λουλέα. Σωστά, Λουλέα, πολύ καλά το είπα. Πολύ καλά, πολύ καλά. Ο Φρέντεκ Φέντεκ ζητά συγγνώμη, ο συνάδελφος δεν μπορούσε να παραστεί. Μου ζήτησε όμως να προβώ σε σύντομη δήλωση, πολύ ενδιαφέρον ταξίδι. Ο Φρέντρικ το οργάνωσε πολύ καλά. Επισκεφθήκαμε το, υβριδικό, το πρόγραμμα Hybrid, είναι ένα πρότυπο ε, χαλιβουργίου πράσινου. Δεν θα παράγει σχεδόν καθόλου αέριο θερμοκηπίου. Αν θέλουμε να απανθρακώσουμε, ε, να μην χρησιμοποιούμε άνθρακα μάλλον, ε, σε αυτό το τομέα, νομίζω ότι αυτό το πρόγραμμα, το hybrid, είναι μια λύση. Και το κέντρο δεδομένων του Facebook, επισκεφθήκαμε, έχει πολύ καλό σύστημα ψήξη φιλικό προ το περιβάλλον. Βέβαια, είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει αυτό στο παγωμένο βορρά τη Σουηδία. Ήταν πάρα πολύ ενδιαφέρον και αυτά έχω να πω για το ταξίδι που κάναμε στο Λούλιο. Πολύ ενδιαφέρουσα συνάντηση, λέει ο πρόεδρο, από καταλαβαίνω. Αποστολή στη Σουηδία. Πρώτη φορά νομίζω που επισκεφθήκαμε τη Σουηδία. Δεν πήγαμε ποτέ πριν. Κάποιες ερωτήσεις, συνάδελφοι. Ορίστε, ο Εντουάρ. Μία ερώτηση για το ιμπριτ. Έχετε κάποιο πρόγραμμα, έχετε... Είναι πολύ μακρύ το χρονικό διάστημα που έχει προταθεί. Μπορεί να επιταχυνθεί το πρόγραμμα για την παραγωγή του καθαρού χάλιβα, να υλοποιηθεί αυτό το πρόγραμμα. Ξέρετε κάτι πάνω σε αυτό. Απάντηση. Το πρόγραμμα Hybrid συνεργασία μεταξύ Φατερφάλ ε, της εταιρείας ενέργειας της LKHB που, της Solvay που είναι χαλιβουργία έχουν δημιουργήσει ένα πρότυπο, ένα εργοστάσιο επίδειξης και στα μέσα του 2020 θα έχουν ένα εργοστάσιο επίδειξης και μέχρι το 2040 ελπίζουν ότι θα λειτουργεί εμπορικά το εργοστάσιο. Θα φτάσουμε στο 2050 σε μηδενικές εκπομπές. Είναι στο μέλλον η προοπτική αυτή, αλλά είναι ένα από τα ελάχιστα έργα, δεν είναι το μοναδικό, που θα μπορεί να παράγει χάλιβα χωρίς εκπομπές αερίων. Το πιο ενδιαφέρον είναι ότι ίσως να μην μπορούν να παράγουν μόνο τελειωμένο προϊόν χάλιβα, αλλά είδος φουγγαριού χάλιβα, ένα συστατικό που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα άλλα χαλιβουργία της Ευρώπης για να παράξουν άλλες μορφές τελικών προϊόντων. Και αυτό θα παράγεται με καθαρή ενέργεια. Δεν θα είναι κάτι σημαντικό μόνο για τη Σουηδική Χαλιβουργία, αλλά για όλη τη χαλιβουργία της ε, Ευρώπης που με αυτή την τεχνολογία θα μπορεί να παράγει χάλιβα χωρίς εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου. Ο κ. Ζητώ συγγνώμη, θα, θα θέσω μια απλούστατη ερώτηση. Ποιο ήταν το μείγμα, η συμμετοχή του υδρογόνου σε αυτό το ε, σιδερένιο ε, σφουγγάρι, τα σιδερένια προϊόντα. Γιατί το υδρογόνο είναι πολύ επιζήμιο ε, κατά τη χρήση χάλιβα για βιομηχανικές ανάγκες, για βιομηχανικούς σκοπούς. Ποιο ήταν το τμήμα του υδρογόνου στο μείγμα. Και εγώ έχω μία ερώτηση. Νέες τεχνολογίες στο χάλιβα, στην παραγωγή χάλιβα. Τι γίνεται με το λιγνίτη στη χρήση τέτοια τεχνολογία γενικά. Υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί το κοκ ή να μην χρησιμοποιηθεί καθόλου το κοκ στο μέλλον για την παραγωγή χάλιβα, καθόλου. Γιατί προς το παρόν δεν φαίνεται ως ρεαλιστικό μέλλον κάτι τέτοιο, να μην χρησιμοποιηθεί καθόλου κόκ στη παραγωγή, αλλά το έχετε σκεφτεί καθόλου. Δυστυχώς δεν είμαι ούτε μηχανικός ούτε επιστήμονας, οπότε δεν μπορώ να σας δώσω μία εκτενή τεχνική απάντηση για την ακριβή χρήση του υδρογόνου. Και δεν πάτε λοιπόν στο Λούλιτ μόνο σας να το εξετάσετε. Θα ήταν πολύ ενδιαφέρουσα εμπειρία σε αυτόν τον βορρά της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Ή να καλέσουμε εκπροσώπους της εταιρεία εδώ στη Βρυξέλλες. Πάντως υπάρχει δυνατότητα χρήση και υδρογόνου και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για να παραχθεί ενέργεια, οπότε θα χρησιμοποιηθεί μεγάλη ποσότητα ενέργειας. Ευτυχώς έχουμε καλό επίπεδο ΑΠΕ, ε, κυρίως από υδροελεκτρική ενέργεια στην ε, Σουηδία. Και φυσικά υπάρχει δυνατότητα να γίνει παραγωγή χωρίς χρήση κόκ. Ε, ελπίζω και στο επόμενο κοινοβούλιο να γίνει αντίστοιχη επίσκεψη στη Σουηδία για την επίσκεψη αυτού του σχεδίου του Ιβριδίου. Θέλω να πω με ταπεινοφροσύνη ότι στόχος της έρευνας αυτής είναι να αποφευθεί η χρήση του κοκ. Ε, γιατί το κόκ είναι καθαρός άνθρακας. Το θέμα είναι να καταργήσουμε πλήρως τον άνθρακα στη χρήση. Γι' αυτό και θα έχουμε μηδενικές ρηπογόνες εκπομπές. Αυτή ήταν μια ε, μικρή ταπεινή παρατήρηση τεχνικού χαρακτήρα. Ναι, το ξέρω. Το ξέρουν. Όποιοι είναι μηχανικοί το γνωρίζουν. Αλλά δεν υπάρχει ακόμη γνωστή τεχνολογία που να μπορεί να στερηθεί τη συμπερίληψη και του κόκ στην παραγωγή. Τελευταία ερώτηση, κύριε Κοχλίτσεκ. Οποιοδήποτε οξύδιο με υδρογόνο μπορεί να περιοριστεί. Πώς θα αποφύγουμε όμως στο σχέδιο να μην μείνουν α, υπολείμματα υδρογόνου. Γι' αυτό ρώτησα. Ποιο είναι το ποσοστό του υδρογόνου που χρησιμοποιείται στο μείγμα του χάλιβα. Αυτό είναι σημαντικό για την περαιτέρω χρήση του προϊόντος. Ποιο είναι το ποσοστό περιεκτικότητα περιεκτικότητας του υδρογόνου στο μείγμα. Εντάξει, αυτό θα το... Θα απαντηθεί στην επόμενη μα επίσκεψη, κοινή επίσκεψη στη Σουηδία. Μάλιστα, συνεχίζουμε. Ενημέρωση σχετικά με τι τρέχουσε διοργανικέ διαπραγματεύσει. Ο συνάδελφο Νίκα θα έρθει σε Κάνα δεκάλεπτο τέταρτο. Ας περάσουμε στο δεύτερο θέμα και θα δώσω το λόγο στον εισηγητή μας, τον κύριο Τζίσουαφ Κρασνοντέμσκι, που θα μας μιλήσει για τη σύσταση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, για τη διαπραγματεύσεις για το θέμα αυτό. Ολοκληρωθήκα στον τρίτο τριμερή διάλογο του Φεβρουαρίου και επετέφθη συμφωνία για μεγάλο τμήμα του κειμένου. Κύριε καθηγητά Κρασοντέμσκι, παρακαλώ, ενημερώστε μας. Ευχαριστώ, κύριε Μπούζεκ. Όπως είπατε, 19 Φεβρουαρίου καταλήξαμε στη συμφωνία. Ήταν ο τρίτος τριμερής διάλογος. 16 Ιανουαρίου, 5 και 19 Φεβρουαρίου ήταν οι τρεις ημερομηνίες. Ε, υπήρξαν διάφορες διαμάχες και συγκρούσεις στην αρχή. Τελικά, στην πορεία των συζητήσεων και των διαπραγματεύσεων, καταφέραμε στον τρίτο τριμερή διάλογο να καταλήξουμε σε συμφωνία μετά από 8 ώρες διαπραγματεύσεις και να καταλήξουμε σε συμφωνία που έτυχε της μεγάλης υποστήριξης των εισηγητών που εκπροσωπούν την πλειοψηφία των ε, πολιτικών παρατάξεων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από αυτά που ζητήσαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πετύχαμε τα εξή σημαντικά. Άμεση ε, διαχείριση του Ταμείου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις περισσότερες περιπτώσεις. Επίσης, ιδιαίτερος ξεχωριστός προπολογισμό προϋπολογισμός για το τεχνολογικό τμήμα, έλλειψη ε, ε ορίων, επίσης για ε, κονδύλια για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και τις μεσαίες κεφαλαιοποίησης επιχειρήσεις. Άλλαξε ε, το σχέδιο κάπως σε σχέση με το ETITP για το άρθρο 7 για τον έλεγχο και τη διαχείριση των σχεδίων. Επίσης, περιορισμένη πρόσβαση σε ό,τι αφορά το είδος των τεχνολογιών και των προϊόντων άμυνας. Άρθρα 11 παράγραφοι 3 και 6. Επιπλέον αποκλείστηκε η χρήση κάποιων κρατικών φορέων ή ε, φορέων που ε, ελέγχονται από το κράτος και που ε, ήταν αντικείμενο κυρώσεων από την Ένωση. Αναφέρεται στην αιτιολογική έκθεση. Επίση, είπαμε ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνα θα στηρίξει τη γενική ανταγωνιστικότητα του ευρωπαϊκού εξοπλιστικού κλάδου. Έτσι το ερμηνεύουν ε, μερικοί, ότι δηλαδή με τα ευρωπαϊκά κονδύλια στηρίζουμε και την ε, αύξηση των εξοπλισμών. Τελικά, μερικά θέματα, όπως το ζήτημα του προγράμματος εργασίας πέρασε στις κατεξιοδότηση πράξης, είναι ιδιαίτερα τα χαρακτηριστικά της αμυντικής βιομηχανίας. Ε, και αυτό έλειφθη υπόψη σε ό,τι αφορά την εφαρμογή του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας από το Συμβούλιο. Πάντως, μαζί με τους συζητητές από το ΕΛ και, την, και τους φιλελεύθερους, συμφωνήσαμε σε αυτή τη λύση ότι το Ταμείο θα, ευχα... εφαρμόζεται μόνο με αιτήσια προγράμματα εργασίας, με κυρίως τη διαδικασία την εκτελεστική, σε αντικατάσταση της προηγούμενης διαδικασίας. Είναι μερική η έχουμε κάποιες εκκρεμότητες οι οποίες θα διαθετηθούν από το επόμενο κοινοβούλιο, όπως το ύψος του προϋπολογισμού, το κρύβος του προϋπολογισμού του, ε, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας, γιατί δεν ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις για το ΠΔΛΤΑΠ και επίσης άρθρο 5 για τα συνδεδεμένα κράτη. Και αυτή είναι η κρεμότητα που θα διαθετηθεί μετά την τελική συμφωνία και με το Ηνωμένο Βασίλειο. Πάντως στο Συμβούλιο δεσμεύθηκε να μην επανέλθει σε θέματα που έκλεισαν στις διαπραγματεύσεις και στις συμβαστικές ε, λύσεις και αύριο 19 Μαρτίου η συμφωνία αυτή θα επιβεβαιωθεί κανονικά στη συνεδρίαση του Συμβουλίου. Να πω για το δικό μου ρόλο καταρχήν να ευχαριστήσω τον, πρωθυπουργό μας, τον πρώην Πρωθυπουργό μας, τον κύριο Μπούζεκ, για τη βοήθεια που μου παρήχε στην τελική και πιο δύσκολη φάση των διαπραγματεύσεων και ως επικεφαλής της διαπραγματευτικής ομάδας προσπάθησα να λάβω υπόψη τις απαιτήσει όλων των πολιτικών ομάδων, ακόμη και αν διαφωνούσα προσωπικά ή αν διαφωνούσε η ομάδα μου με τις απόψεις άλλων πολιτικών ομάδων. Εγώ προσπάθησα να εκπροσωπήσω το σύνολο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και να κάνω μια ρεαλιστική και αντικειμενική ε, εκτίμηση της κατάστασης. Και την επόμενη Δευτέρα θα ψηφίσουμε στην Ήτρε την Επιτροπή μας και θα πάει το θέμα στην Ολομέλεια της 4 η Απριλίου. Ελπίζω ότι οι συνάδελφοι και από τις ομάδες που δεν έμειναν απόλυτα οικονοποιημένες να αναγνωρίσουν παρόλα αυτά την επιτυχία που σημειώσαμε σε πολλά επιμέρους σημεία για το θέμα αυτό που ήταν σημαντικά στις διαπραγματεύσεις και Ελπίζω να συγκεντρώσουμε την ε, απαραίτητη πλειοψηφία και να επιβεβαιώσουμε τη συμφωνία αυτή με το Συμβούλιο στον Τριμερή Διάλογο. Σας ευχαριστούμε κύριε Κρασνοντέμψη για την ενημέρωση και για την έκβαση των διαπραγματεύσεων. Όπως είπατε, η ψηφοφορία θα γίνει σε μια εβδομάδα εδώ στην Ήτρε. Ποιο θέλει το λόγο, παρακαλώ. Ο κύριος Μαχτά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και ευχαριστώ και τον συνάδελφο Κρασνοντέμσκι τον εισηγητή μας για την ενημέρωση. Όπως είπε και στο τέλος υπάρχουν σημεία με τα οποία διαφωνούμε κάθετα, παρόλα αυτά αναγνωρίζουμε το έργο του. Τα του Κέσσερο στο Κέσσερι. Ο εισηγητής έβαλα τα δυνατά του και ανταπεξήλθα όπως μπορούσε στην εντολή που του είχαμε δώσει. Μπορεί να μην είμαστε απόλυτα ικανοποιημένοι, πάντως αγνωρίζουμε την προσπάθειά του. Ήταν η πρώτη εμπειρία που είχα σε διαπραγματεύσει με το Συμβούλιο και πρώτη φορά είδα να μου λέει ο συνομιλητής ότι δεν έχω ε, εντολή για τίποτα. Τι διαπραγματευτική τακτική είναι αυτή. Ε, είναι σαν να μην είχε καμία εξουσία εκπρόσωπος του Συμβουλίου. Μας έλεγε συνέχεια: Δεν μπορώ να δώσω λευκό επιταγή, θα με επιπλήξουν. Αυτά είναι αερολογίες. Γνωρίζουμε αυτές τις διαπραγματευτικές τακτικές. Ξέρω ότι περί τακτικής πρόκειται και δεν θα ε, έπρεπε να πέσουμε σε αυτή την παγίδα. Επί της ουσίας τώρα, η δέσμευση του Συμβουλίου, η περίφημη επιστολή που θα μα στείλει το Συμβούλιο και που φαίνεται θα δίνει εγγύηση ότι δεν πρόκειται να αφισβητηθούν τα διαπραγματεύοντα. Αυτό, αυτή η επιστολή του Συμβουλίου όμω είναι σαν το τέρα του Λοχνέ. Όλοι μιλάνε γι' αυτό, αλλά κανένα δεν το έχει δει. Ποιο μπορεί να είναι το περιεχόμενο τη επιστολή. Το μόνο που μπορεί να κάνει το Συμβούλιο είναι να λάβει γνώση του αποτελέσματο τη διαπραγμάτευση. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να δώσει εχέγγυα η εγγυήση ότι δεν θα επανέλθει στα θέματα αυτά. Ουσιαστικά υπογράφουμε λευκό επιταγή, γιατί δεν θα έχουμε κατεξοδότηση πράξη. Οπότε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σχεδόν... Εντάξει, εγώ, εμένα στα παλιά μου τα παπούτσια, γιατί δεν θα ξαναέρθω εδώ στο κοινοβούλιο. Αλλά το επόμενο κοινοβούλιο θα έχει καθόλου δυνατότητα να παρεύει στο πρόγραμμα εργασιών. Και 13 δισεκατομμύρια ευρώ είναι ο υποθετικό προπολογισμό. Αλλά δεν έχει κλείσει το θέμα. Και το βασικό εδώ είναι το οικονομικό θέμα. Θα είναι 13 5, 7 ποιο θα είναι το τελικό ποσό προπολογισμό του Ταμείου Άμυνα. Γιατί δεν γνωρίζουμε το ύψο του ποσού. Μιλήσατε για το άρθρο 5 ή επιλέξιμες μεσοντότητες. Και εκεί διαφωνούμε. Επίσης, για τα θανατηφόρα όπλα. Επίσης, συμμετείχα στην αποστολή επιστολή στον πρόεδρο Ταγιάννη, στη διάσκεψη των προέδρων και σε εσά κύριε Μπούζεκ. Ήσταν ένας από τους παραλήπτη τη αποστολή. Και δεν ξέρουμε αν υπάρχει συμφωνία, γιατί η διάσκεψη των Προέδρων δεν έλαβε ακόμη θέση. Και υπενθυμίζω ότι η θέση των Προέδρων ήταν από την αρχή ότι δεν θα συμφωνήσουμε ή δεν θα κυρώσουμε μια συμφωνία αν απορριφθεί το αίτημά μα για την κατεξοδότηση πράξη. Και αυτό ήταν από την αρχή η θέση του Συμβουλίου ότι αποκλείεται, ξεχάστε τις κατεξοδότηση πράξη. Εμείς που είμαστε εκπρόσωποι των Ευρωπαίων πολιτών έχουμε μείνει με σταυρωμένα χέρια. Μα έχουν δέσει τα χέρια μάλλον με αυτόν τον αποκλεισμό των κατεξοδότησε πράξη, με την αποκλεισμό των πράξη. Διάβασα στι εφημερίδες ε, την περασμένη εβδομάδα ότι η πολωνική κυβέρνηση ήθελε να ε, ενισχύσει τους εξοπλισμούς και προέβλεπε προϋπολογισμό 40 δισεκατομμύρια ευρώ για να ενισχύσει τους εξοπλισμούς και την ασπίδα προστασίας. Σε ποιο θα κάνει παραγγελία σας δίνω μια πιθανή πρόβλεψη. Στους Αμερικανούς θα παραγγείλει πολεμικούς εξοπλισμούς η Πολωνία μάλλον. Κύριε Γκροστέτ. Ε, λυπάμαι, μόλις έφτασα. Το τρένο μου είχε μεγάλη καθυστέρηση από το Παρίσι. Θα προτιμούσα να είμαι παρούσα και να, ακούσα το, να ακούσω τον εισηγητή. Ξέρετε πολύ καλά την υπόθεση κύριε Πρόεδρε. Να σε ευχαριστήσω για το ρόλο που παίξατε έναντι του Σιγητού για να βοηθήσετε την επίτευξη συμφωνίας. Δεν ήταν απλά τα πράγματα. Ήταν περίπλοκα. Εύκολο να επικρίνει κανείς. Πάντα υπάρχουν κάποιες αποφάσεις που θα θέλαμε να είναι διαφορετικές. Πρέπει να γνωρίζετε ότι πρόκειται περί θέματος ε, ιδιαίτερου. Η άμυνα σχετίζεται με την κυριαρχία των κρατών μέλων και αυτό εξηγεί ότι έπρεπε να δεχθούμε κάποια πράγματα, διότι επρόκειτο περί ζητήματος ιδιαίτερος ευαισθητού. Αν θέλαμε μια συμφωνία με το Συμβούλιο, έπρεπε να λάβουμε υπόψη αυτό το θέμα που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητο, διότι άπτεται τις κυριαρχίες των κρατών μελών. Δεν θα αναφερθώ στις λεπτομέρειες, υποστηρίζω προφανώς την επιτευχθήσα συμφωνία αυτή που πέτυχε ο εισηγητής μετά από πολλές ώρες συζητήσεων και διαπραγματεύσεων. Δεν ήταν πάντα απλά τα πράγματα. Απέναντί μας είχαμε ένα συμβούλιο που είχαμε το συνέστημα σε κάποια φάση ότι δεν ήταν καλά προετοιμασμένο. Πιστεύω ότι πρέπει πράγματι να υποστηρίξουμε αυτή τη συμφωνία. Ελπίζω ότι το επόμενο κοινοβούλιο στα πλαίσια του προπολογισμού θα υπερασπιστεί τις οικονομικές δεσμεύσεις που προβλέπονται, διότι είναι απαραίτητες. Συμφωνώ με τον συνάδελφο Εντουάρ Θα πρέπει τα κράτη-μέλη να παίξουν το παιχνίδι τους. Θα πρέπει να κινηθούν. Θα συμμετάσχουν, πιστεύω, διότι σε επιχειρήσεις όπως αυτή, αυτό που θα χρηματοδοτηθεί και θα υποστηριχθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τα προγράμματα θα είναι εκείνα στα οποία θέλουν να συμμετάσχουν τα κράτη-μέλη. Αν θα συμμετάσχουν οικονομικά, σημαίνει ότι θα συμμετάσχουν αναγκαστικά αγοράζοντας, αποκτώντας αυτό που θα είναι προϊόν του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας. Θέλω να υποστηρίξω τη συμφωνία. Στηρίζει το ΕΛΚ τη συμφωνία στηρίζει αυτές τις διαπραγματεύσεις δεν ήταν καθόλου εύκολες. Και τελικά καταλήξαμε σε αυτό που είχε αποφασιστεί στο πρώτο σχέδιο για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας 2019-2020 γυρίσαμε στα βασικά, στα θεμελιώδη. Είναι καλό. Θα πρέπει λοιπόν να υποστηρίξουμε αυτή τη συμφωνία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Καθηγητά, θέλετε να δευτερολογήσετε για να συνοψίσετε. Να θα μιλήσω αγγλικά αυτή τη φορά. Καταρχάς λοιπόν, να τονίσω ότι κάθε φορά που καταλήγουμε σε ένα συμβιβασμό δεν σημαίνει πως όλοι μένουν ικανοποιημένοι. Και σίγουρα υπάρχουν επιθυμίες που δεν εκπληρώθηκαν τώρα. Σε ό,τι αφορά τη δέσμευση των κρατών μελών, να σας πω πως αύριο, 19 Μαρτίου, θα λάβει χώρα μία συνάντηση και είμαστε σίγουροι πως η επιστολή θα σταλεί τότε. Και θα έχουμε τη γραπτή δέσμευση του Συμβουλίου στη συμφωνία αυτή. Να πω επίσης ότι, όπως είπε και η κυρία Γκροστέτ, ο ρόλος των κρατών μελών είναι ιδιαίτερα ενισχυμένος εδώ. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα αυτό για τα κρατημέλη, γι' αυτό και μπορέσαμε να δεχτούμε τις εκτελεστικές αυτές πράξεις ως ε, τον τρόπο που θα επιληθεί το πρόβλημα αυτό. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη, έγινε δεκτή η ίδια λύση. Γι' αυτό λοιπόν δεν νομίζω πως υπάρχει κάτι καινούργιο εδώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ήταν καλοδεχούμενη η στήριξή σας. Σας ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Έλλερ θέλει να προσθέσει κάτι. Με συγχωρείτε κύριε Έλερα, αλλά είχα την εντύπωση ότι ζητήσατε το λόγο για το πρόγραμμα Ορίζοντας Ευρώπη. Ε, σας παρακαλώ, ναι, ε, τοποθετηθείτε. Θα ήθελα να αναφερθώ και εγώ στους ε, προβληματισμούς που είχε ο κύριος ε, Μαρτάν. Χρειάζεται να παρασχεθούν ορισμένες διασφαλίσεις για τα ταμεία που δεν θα απορροφηθούν πλήρως, όμως να πω πως δεν είναι πρώτη φορά που η κρίση του Κοινοβουλίου εξαρτάται από την απόφαση του Συμβουλίου για τη μορφή της συμφωνίας που θα είναι δεσμευτική και τις δύο πλευρές. Ε, δεν έχει γίνει λοιπόν πρώτη φορά αυτό. Να σας υπενθυμίσω ότι συνηθίζεται στις διαπραγματεύσεις για το πολίτες δημοσιονομικό πλαίσιο να λάβουμε έναν κλειστό δημοσιονομικό φάκελο, ο οποίος είχε ήδη διαπραγματευτεί. Και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε τη δυνατότητα ή να περικόψει ή να υπερβεί τον προϋπολογισμό χωρίς όμως να έχει αυτό επιπτώσει στην ουσία της πρότασης. Εάν λοιπόν εμείς λάβουμε τη διασφάλιση πως ε, θα δεσμευτεί το Συμβούλιο, θα συμβεί για πρώτη φορά οι διαπραγματεύσεις για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο να στηρίζονται σε μια βάση. Διότι στο παρελθόν οι διαπραγματεύσεις αυτές ήταν στην ουσία μια αφηρημένη συζήτηση για τον προπολογισμό. Μετά παίρναμε το φάκελο με τα στοιχεία και αυτό ήταν. Γι' αυτό θεωρώ πως από τεχνικής άποψης ε, θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο να έχουμε αυτές τις διασφαλίσεις ότι στις ε, διαπραγματεύσεις για το που δε που θα ξέρουμε ε, περί τίνος πρόκειται και γιατί πράγμα διαπραγματευόμαστε. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν μας μένει χρόνο διότι, χρόνος διότι έχουμε τέσσερα ακόμα θέματα να συζητήσουμε. Τέσσερις ενημερώσεις πριν τη συνάντηση των συντονιστών. Να προσθέσω όμως και κάτι τελευταίο. Ο κύριος συζητητής αναφέρθηκε στη διευκόλυνση συνδέοντας την Ευρώπη. Θεωρώ πως συνδέεται και με την έκθεση της ε, κυρίας Γκροστέτ. σχετικά με την ε, ανάπτυξη της εξοπλιστικής βιομηχανίας. Υπάρχουν πάρα πολλέ ομοιότητε εδώ. Παρ' όλα αυτά, δείξαμε την αντίδρασή μας και τι αντιρρήσει μας για να μην είναι τόσο εύκολα τα πράγματα για το Συμβούλιο. Κύριε Μαρτάν, θέλετε να πάρετε το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Μισό λεπτό μα. 30 δευτερόλεπτα για αυτά που είπε ο Σέλλο. Συμφωνώ με αυτό. Αλλά δεν διαμαρτύρομαι γι' αυτό. Ξέρουμε ότι άλλοι θα διαπραγματευτούν. Αλλά Στη, στη διάσκεψη των Προέδρων, οι Πρόεδροι έλαβαν απόφαση. Είπαν ότι να αρνηθούν την συμφωνία αν δεν υπάρχει κατεξουδότηση πράξη. Αυτό συγκρατώ. Δεν ξέρω τι αποφάσισε ή θα αποφασίσει την πέντε έξω των Προέδρων. Δέχτηκα να υποβληθεί σε ψηφοφορία η θα αποφασισει την πεντε του των προεδρων δεχτηκαν να υποβληθει σε ψηφοφορια η συμφωνια Επ' αυτού έχω το πρόβλημα, ότι ανοίγουμε ένα κενό για τις άλλες διαπραγματεύσει, Προηγούμενο δημιουργούμε. Ευχαριστώ, όπως ξέρετε. Προσθέσαμε δύο νέα σημεία στην Ευρωπαϊκή, στην ημερήσια μας διάταξη, το Ευρωπαϊκό Κέντρο Έρευνα και Ικανοτήτων Ασφάλεια στον Κυβερνοχώρο. Μα ενημέρωσε γι' αυτό η κυρία Γιουλία Ρέντα πριν από λίγο. Και τώρα ο κύριο Λεβαντόφσκι θα μα ενημερώσει για τι ευρωπαϊκέ στατιστικέ για τι επιχειρήσει. 14 ε, Μαρτίου έγινε ο σχετικό τριμερή διάλογο στο Στρασβούργο. Επιτυχημένο ήταν ο διάλογο και καταλήξαμε σε προσωρινή συμφωνία με το Συμβούλιο για αυτό το πολύ τεχνικό θέμα, τον Ευρωπαϊκό Στατιστικό για τις Επιχειρήσεις. Τεχνικό και περίπλοκο. Μία δεκαετία ολόκληρη χρειάστηκε για να καταλήξουμε σε συμφωνία για το θέμα αυτό των Ευρωπαϊκών Στατιστικών για τις Επιχειρήσεις. Σε ένα πολύ μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον που επεκτάθηκε και στις ε, υπηρεσίες, στο διεθνές εμπόριο, στις ε, τεχνολογίες πληροφορίες και επικοινωνίες. Πάντως, Πραγματικά συνιστούμε απλούστευση γιατί αντικαθιστούμε δέκα νομικές πράξεις με έναν και μόνο κανονισμό. Αυτό και αν είναι απλοποίηση και έτσι μειώνουμε και τη γραφειοκρατία με την αντικατάσταση αυτών των 10 νομοθετικών πράξεων από μία. Είχαμε και κατακαιρματισμό. Θέλησαμε να μειώσουμε εκτός από τη γραφειοκρατία και το κόστος, κυρίως για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και να εξασφαλίσουμε και την εμπιστευτικότητα στο θέμα των στατιστικών. Μερικές ε, θέσεις του Συμβουλίου ήταν ιδιαίτερα άκαμπτες. Τελικά καταφέραμε να τις κάμψουμε κάπως, να τις καταστήσουμε πιο ελαστικές, λαμβάνοντας υπόψη και το μεταβαλλόμενο επιχειρηματικό περιβάλλον και κλίμα. Έχουμε κάποιους νέου δείκτες στα θέματα της χρηματοδότησης και των κλιματικών αλλαγών, που θα είναι το αντικείμενο πιλωτικών μελετών. Πάντω είχαμε την πρόθεση να τι περιλάβουμε στο θέμα αυτό. Ευχαριστώ τους και οδησηγητές, την κυρία Κούπουλα Νάτρη από το S&D, τον Μάρικ από το ECR, Τελίτσκα, Λόπες Βερμέχο, Κάπελ και ούτω καθεξής. Και ευχαριστώ και τους συμβούλους μας, την Κάσια, τον Κλάους και φυσικά τον Τόμεκ και την Τατιάνα μετά από 10 χρόνια καταφέραμε να διεκπαιρεώσουμε αισίως ε, την προσωρινή συμφωνία. Την επόμενη Δευτέρα θα ψηφίσουμε στην Επιτροπή μας Ήτρε, προκειμένου να διαβιβάσουμε το ζήτημα στην Ολομέλεια του Στρασβούργου την τελευταία του Απριλίου. Ευχαριστώ. Άλλος κανείς? Θέλει το λόγο. Όχι. Ευχαριστούμε κύριε Λεβαντόφσκι για την σύντομη και περικτική σας ενημέρωση και να πάμε τώρα στο σημείο 10, το ορίζον Ευρώπη, εδώ έχουμε δύο συνεισηγητές, τον κύριο Νταν Νίκα και τον κύριο Κρίστιαν Έλερ. Παρακαλώ, ενημερώστε μας. Τι γίνεται με το πρόγραμμα Ορίζον Ευρώπη. Είναι πολύ περίπλοκο το θέμα. Την περασμένη πέμπτη λοιπόν καταφέραμε να ολοκληρώσουμε τη συμφωνία όμως κατέστη προφανές ότι η δέσμη μέτρων την οποία διαπραγματευτήκαμε ήταν δύσκολο να ε, γίνει αποδεκτή από όλους. Τώρα, οι προκλήσεις εδώ έχουν να κάνουν με το ότι από τη μία πρόκειται για δύο θέματα, ε, στα οποία υπάρχει η διαδικασία συναπόφασης και συμμετέχει κομισιόν και, και υπάρχει και η τρίτη δέσμη μέτρων για τον στρατηγικό σχεδιασμό που δεν βρισκόταν ούτε στον, ε, στο φάκελο αυτό ούτε στον κανονισμό. Οπότε λοιπόν που είναι η νομική βάση. Η θέση του Κοινοβουλίου είχε ως εξή. Ο στρατηγικός σχεδιασμός είτε θα είναι πράξη κατά εξουσιοδότηση εφόσον δεν βρίσκεται σε καμία από τις δύο προτάσεις είτε θα πρέπει να αναπαιμφθεί στους, ε, στα δύο θέματα συναπόφασης ή στον κανονισμό. Ίσως καταφέρουμε να βρούμε μια λύση, διότι το Συμβούλιο ήταν πρόθυμο να επανεισαγαγεί τον στρατηγικό σχεδιασμό στον κανονισμό και οι εκκρεμότητες έχουν να κάνουν με επιτροπολογία και με τις εκτελεστικές πράξεις. Γι' αυτό λοιπόν ε, Νομίζω πως θα καταφέρουμε αυτό που θέλουμε, στην ουσία πράξεις κατά εξουσιοδότηση ω θέση του Κοινοβουλίου, αλλά το αποτέλεσμα των διαπραγματεύσεων ήταν να επανεισεχθεί στον ε, φάκελο που είναι αντικείμενο συναπόφασης και το Κοινοβούλιο να ενισχύσει τη θέση του, διατηρώντα αυτέ τι πράξει κατά εξουσιοδότηση. Στην ουσία τώρα, για το δεύτερο θέμα, για την έκθεσή μου, το πρόβλημα που παρουσιάστηκε είναι ότι το Συμβούλιο αμφισβήτησε ε, επίσημα την ε, νομική βάση. Γι' αυτό λοιπόν καταλήξαμε σε μια διελκυστίνδα. Θέλουμε δηλαδή να ξεκινήσουν επίσημα διαπραγματεύσεις ενώ συζητούμε ακόμα τα δύο θέματα και ταυτόχρονα το Κοινοβούλιο να ε, καταθέσει μια συμβαστική πρόταση που θα καλύπτει όλες τις ε, πτυχές, μια που υπάρχει αυτή η διασύνδεση. Ή δεύτερον, να συνεχίσουν οι διαπραγματεύσεις και μετά να δούμε τι θα κάνουμε. Α, κατά πάσα πιθανότητα στον τελευταίο τριμερή διάλογο θα καταλήξουμε σε μια θέση για την νομική βάση για τα δύο αυτά θέματα και για το στρατηγικό σχεδιασμό και έπειτα ουσιαστικά να πω ότι το 70% περίπου των ε, θέσεων του Κοινοβουλίου έγιναν αμέσω δεκτέ από το Συμβούλιο, το 1 τέταρτο όχι. Και τα θέματα που δεν έγιναν δεκτά είχαν να κάνουν με την ε, διεύρυνση της δέσμης μέτρων, με διάφορα στοιχεία σχετικά με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και με ε, το γεγονός ότι το Συμβούλιο θέλει να εξαιρέσει την κινητικότητα και να εξεταστεί αυτή μόνη της. Στην ουσία, οι συμβιβασμοί ήταν αρκετά ικανοποιητικοί. Καταφέραμε λοιπόν να φτάσουμε σε αποτελέσματα. Νομίζω ο τριμερής διάλογος που θα ακολουθήσει θα είναι ο 7 αύριο στις 5.30 το απόγευμα. Αυτή λοιπόν είναι μια πολύ γενική εικόνα της κατάστασης και του που βρισκόμαστε. Και αν ενδιαφέρει τους συναθέλφους ε, να πω ότι συζητήθηκε και το θέμα της ε, παραγωγής διοξιδίου του άνθρακα από τη Χαλιβουργία, όπου προτάθηκε από το Συμβούλιο μια γενικότερη παρέμβαση η οποία προβλέπει να βγει ο άνθρακας από την καύση και αυτό είναι μια πρόκληση σε ουσιαστικούς όρους. Βέβαια αυτή η πρόταση δεν έφτασε ποτέ πέρα από το πιλωτικό στάδιο και τώρα το θέμα είναι τι θα κάνουμε με τη χρηματοδότηση, πού θα βρεθούν χρήματα. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο ενδιαφέρει πάρα πολύ το Κοινοβούλιο διότι ενδιαφέρει πάρα πολύ και την ε, βιομηχανία και το διάλογο που εκτελήσεται αυτήν την ε, περίοδο και το Συμβούλιο φαίνεται να αποδέχεται τις ε, θέσεις μας. Σας ευχαριστώ πολύ. Υπάρχουν ερωτήσεις ή σχόλια. Δεν βλέπω κάτι τέτοιο, οπότε μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο σημείο. 12. Θέσπιση του Διαστημικού Προγράμματος της Ένωσης και του Οργανισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το Διαστημικό Πρόγραμμα. Η είναι ο Μασιμιλιάνο Σαλίνη. Ο δεύτερος τριμερής διάλογος έλαβε χώρα στις 20 ε, Φεβρουαρίου και θα δώσω αμέσω το λόγο στον εισηγητή για να μας ενημερώσει. Ευχαριστώ πολύ, θα μιλήσω τη γλώσσα μου. Η κατάσταση με τον τελευταίο τριμερή διάλογο επελήθη, είχαμε δύο τριμερείς διαλόγους, ε, έγινε διάφορες πολυάριθμες τεχνικής φύσης συναντήσεις, η απόφαση είναι αρκετά ικανοποιητική, δεν θα επεσέλθω στις κατεξοδότηση αλλά σε όλο το θέμα που αφορά το γενικό πακέτο του πολιτού δημοσιονομικού πλαισίου, διότι είναι πολύ παρόμοια τα επιχειρήματα με αυτά που είπαν οι συνάδελφοι, αλλά θα επικεντρωθώ επί των διαπραγματεύσεων που ολοκληρώθηκαν. Όσον αφορά τη διακυβέρνηση, ένα τελευταίο σημείο πάρα πολύ νομική φύσεως θα έλεγα, αλλά που έχει συνέπειες όσον αφορά τη ζωή των υπηρεσιών που ετέθη τον τελευταίο τριμερή διάλογο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και είπε συγκεκριμένα στο θέμα της υποανάθεσης βρήκαμε μία σωστή λύση να αλλάξουμε το περιεχόμενο χωρίς να συγκληθεί, η νέο τριμερής διάλογος. Είμαι πολύ ικανοποιημένος από αυτή την απόφαση όπου το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο πέτυχαν συμφωνία και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συνεργάστηκε για να καθοριστεί το τεχνικό περιεχόμενο θα γίνουν στην Ήτρε και στην Ολομέλεια θα πάμε τον Απρίλιο. Ως αφορά φάση των συζητήσεων και για τις διάφορες προσπάθειες που έγιναν, ευχαριστώ τη γραμματεία και τη γραμματεία του ε, κόμματός μου, του συναδέλφου ευχαριστώ επίσης, τους κοιόδης εισηγητές. Πιστεύω ότι θέσαμε τη βάση μια, μια τέλεια, μια πάρα πολύ καλή κατάληξη των συνομιλίων. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ συνάδελφε. Δεν μπορώ να συγχαρώ όλους σας για τα αποτελέσματα των τριμερών διαλόγων. Είχαμε πολλούς τριμερείς διαλόγους, έχουμε πολλούς στην Επιτροπή, πέντε ολοκληρώθηκαν, δύο από αυτούς τους διαλόγους συνεχίζονται, αλλά πάρα πολλούς διαλόγους. Αν συγκρίνουμε με τις άλλες επιτροπές, ευχαριστώ πάρα πολύ συνάδελφε, ζητάει κάποιος το λόγο για αυτό το θέμα, διαστημική πολιτική διαστημικό πρόγραμμα. Δεν ζητάει κανεί το λόγο. Επόμενο σημείο. Ένα βιρκούνεν. Η δημιουργία του μέσου για διασύνδεση της Ευρώπης, Connecting Europe Facility. Έχουμε, είμαστε αρμόδια επιτροπή μαζί με την Επιτροπή Μεταφορών και ο τελευταίος τιμερής διάλογος έλαβε χώρα στις 7 Μαρτίου. Η ε, Χάνα έστειλε κάποιες συμφ... ε, Η συμφωνία που επετεύθη καλύπτει όλο το κείμενο εκτός από τα στοιχεία στο, τετραγωνίδιο του Συμβουλίου ε, στοιχεία, τρίτες χώρες, ε, τα θέματα εκείνης διαχείρισης. Η ε, Κορεπέρ θα, το συζήτησε 25 Μαρτίου θα ψηφίσουμε ψηφιακό τομέα, σημαντικά. Ο τριμερής διάλογος κατέχει αποτελέσματα βάσει της εκθέσεως του Κοινοβουλίου για τον καθορισμό των προγραμμάτων κοινο, κοινού συμφέροντος και εκεί αυτό κατέστη πιο σαφές για τα διάφορα ψηφιακά προγράμματα και στον ενεργειακό τομέα επετέφθησαν καλοί συμβιβασμοί με το ποσοστό ανανοσίμων πηγών ενέργειας και ο μηχανισμός για τη χρηματοδότηση αυτό και αναθεώρηση του, των διαευρωπαϊκών δικτύων. Αυτά είναι τα πιο σημαντικά θέματα. Αυτά μας λέει η κυρία Σιγήτρια ενημερωτικά. Η κυρία Βιρκούνεν. Η αντιπροσωπεία του, της Ήτρες στο Ισραήλ. Ο κύριος Ρούμπικ ήταν επικεφαλής. Στην επόμενη συνεδρίαση θα γίνει ενημέρωση. Ο κύριος Ρούμπικ αναμενόταν να έρθει, αλλά δεν ήρθε, δεν είναι παρόν. Η επόμενη συνεδρίαση 25 Μαρτίου του 2019 στο Στρασβούργο. Σε μια εβδομάδα λοιπόν, Δευτέρα στο Στρασβούργο, 8.30. Στις 8.30, πολύ αργά. Θα είσαστε παρόντες όλοι και θα έχουμε πολλές ψηφοφορίες από ό,τι ξέρω. Λίγο περισσότερες ψηφοφορίες από ό,τι σήμερα. Και τώρα θα γίνει συνεδρία των συντονιστών σε μερικά λεπτά. Ευχαριστώ πάρα πολύ τα μέλη της Επιτροπής Ήτρε και τους βοηθούς συμβούλους. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας και θα συνεδριάσουμε και κλεισμένων των θυρών συνεδρίσεις των συντονιστών. Γεια σας.